Bien, mes chers collègues, je vous invite à regagner votre place, s'il vous plaît. Παρακαλώ καθίστε ξανά. Έχουμε μια ιδιαίτερα φορτωμένη μερίσια διάταξη. Σήμερα το απόγευμα λαμβάνει χώρα ε, συνεδρίαση έρωτα αποκρίσεων στο πλαίσιο της ε, ε, κοινής συνάντησης Econ Budget, Budge, εγώ δεν θα είμαι παρόν, δυστυχώς δεν μπορώ. Ευχαριστώ τον κύριο Γκάλερ που θα προεδρεύσει στη θέση μου σε συνεργασία με τον κύριο Γκουαλτιέρη. Ξεκινάμε λοιπόν. Ποιες είναι οι αποφάσεις που πήραμε οι συντονιστές. Αποφασίσαμε καταρχήν να μην υποβάλουμε έκθεση γνωμοδότησης για την πρόταση απόφαση Συμβουλίου για τη δημιουργία της Επιτροπής Απασχόλησης και καταργεί την απόφαση για τη ε, δημιουργία της Επιτροπής Κοινωνικής Ασφάλειας. Επίσης ε, κατανείμαμε τις ε, εκθέσεις, μία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στον κύριο Γκέρεντς των ε, φιλελεύθερων μια γνωμοδότηση για την πρόταση ρύθμισης σχέδιο πρωτοβουλίας, πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, πρωτοβουλία, ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ε, και πάλι φιλελεύθερη επί τη βάση του κανόνα 53 συν και εγώ θα είμαι συγητής έκθεση για το, το Άρθρο 23 του κοινού κανονισμού, ε, εφαρμοστικές διατάξεις, ε, θα αναλάβει το ΕΛΚ, θα μας ενημερώσει για τον εισηγητή τις επόμενες μέρες. Οι συντονιστές της 11 η Φεβρουαρίου ε, αποφάσισε για το σεμινέο της 31ης Μαρτίου επιβεβαιώσαμε τον κατάλογο των εξωτερικών ε, συμμετεχόντων ε, του συντονιστή και αυτού που θα λάβουν το λόγο ε, για το κάθε ένα από τα πάνελς. Σε ό,τι αφορά την αποστολή στην Ουκρανία που θα γίνει στις 17 και 18 Μαρτίου η ομάδα θα περιλαμβάνει τρεις από το ΕΛΚ, δύο από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες και έναν από τους φιλελεύθερους. Σε ό,τι αφορά τις ακροάσεις. Πέραν των κοινών ακροάσεων που έχουν ήδη ε, αποφασιστεί, για παράδειγμα αυτή που έγινε με τη ΣΕΝΤΕ για την πολιτική ασφάλειας και άμυνας, στις 21 Ιανουαρίου είχαμε επίσης μία κόμμα κοινή με την ε, ΕΚΟΝ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων θα λάβει χώρα την επόμενη Δευτέρα 2 Μαρτίου μία τρίτη με τον, ε, τον ελέγχο του προπολογισμού για τους ιδίους πόρους θα λάβει χώρα στις 5 Μαΐου και οι υπόλοιπε θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του 2015 μία για τον κύκλο πληρωμών και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, την προχρηματοδότηση, τις προκαταβολές τον, και την τελική καθάριση, πώς όλα αυτά οργανώνονται, πώς οργανώνεται αυτή η αλυσίδα πληρωμών και ποιες είναι οι διαδικασίες. Δεν έχουμε ακόμα ημερομηνία για αυτήν την ακρόαση. Για το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων θέλουμε να δούμε ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση, να δούμε πώς γίνεται ε, η δέσμευση των ποιώσεων 2014-2015 και θα λάβει χώρα στην αρχή του 2016 τελικά. Σε ό,τι αφορά τις ε, συναντήσεις των συντονιστών για το πρώτο εξάμεινο του 2015. Εγκρίναμε το χρονοδιάγραμμα, καθώς επίσης και το χρονοδιάγραμμα των διαφόρων φάσεων έγκρισης του προσχεδίου προπολογισμού 2016. <coughs> Για το 2016 οι συντονιστές ενέκριναν το χρονοδιάγραμμα για την έκθεση Φερνάντες. Σε ό,τι αφορά το πολιετές δημοσιονομικό, ε, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, αποφασίσαμε να εκδώσουμε έκθεση για την ε, έγκριση, ε, για τη συνένεση, report on consent, και το πολιτικό μήνυμα θα έρθει όταν εξεταστεί και ψηφιστεί ο διορθωτικό, το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού, το DAB 1. Ε, Σε τη φορά το πρόγραμμα επενδύσεων, οι συντονιστές ενέκριναν το χρονοδιάγραμμα των διαφορετικών συναντήσεων που καθορίζεται από κοινού με την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Είναι ιδιαίτερα πιεστική και Για τις πληρωμές. Οι συντονιστές αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια ομάδα ad hoc για να προετοιμάσει και να διαπραγματευθεί τους όρους του ε, προγράμματος ε, καθάρισης των ε, εκκρεμών των λογαριασμών για τα έτη 2014-2015-2016. Οι συγητές θα συμμετάσχουν σε αυτή την ομάδα και ο πρόεδρος επίσης. Στις 23 Φεβρουαρίου συζητήσαμε την Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα οι συντονιστές ανέθεσαν στον Πρόεδρο να έρθει σε επαφή με τους Προέδρους της ε, ε, ΕΚΟΝ και της Επιτροπής Απασχόλησης για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα από αυτή τη βδομάδα. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη. Ε, εγώ που την παρακολούθησα ως βουλευτής φέτος και ε, ως ευρωβουλευτής φέτος και ως εθνικός βουλευτής προηγούμενες χρονιές νομίζω ότι μπορούμε να τη βελτιώσουμε και χρειάζεται να τη βελτιώσουμε αν θέλουμε να τη διατηρήσουμε. Σε ό,τι αφορά τις ε, μήνυ ολομέλειες. Ε, επιθυμούμε, είπαμε, να εξακολουθούν να γίνονται ψηφοφορίε εδώ στι μήνυ ολομέλη τη. Έχουμε κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να ψηφίζονται επιγόντω. Ε, για να μπαίνουν σε ισχύ. Οπότε οι συντονιστές των διαφορετικών ομάδων ειδοποιήθηκαν έτσι ώστε να πιέσουμε οι, οι ψηφοφορίες και οι οι ολομέλειες να διατηρηθούν στις ε, Βρυξέλλες. Αλλιώς θα καθυστερούμε και θα μας κατηγορούν ότι αδρανούμε. Αυτά σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις των συντονιστών. Πήρε και τα πρακτικά της 5ης Φεβρουαρίου, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσεις. Όχι, εγκρίνουμε τα πρακτικά της 5ης Φεβρουαρίου. Περνάμε στο σημείο 4. Με τη βάση του κανόνα 59 το Κοινοβούλιο ψηφίζει επί του συνόλου των ψηφισμάτων που περιλαμβάνουν μια δήλωση μόνο, μια δήλωση που αναφέρει αν το Κοινοβούλιο δέχεται ή α, απορρίπτει ή τροποποιεί την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ε, η, η προθεσμία είναι 11 Μαρτίου. Ο ο κανόνας 99.1 αναφέρει ότι ε, οι προτάσεις ε, μπορούν να γίνουν δεκτές μόνο ε, για να αμφισβητηθεί και να ανατραπεί αυτό προτείνει ο συγητής. Ο λόγος στην κυρία Τομά. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως, με τον κύριο Όλμπριχτ ε, είμαστε εισηγητές, αλλά δυστυχώς ε, δεν μπορεί να παραβρεθεί ο κύριος Όλμπριτ. Αλλά συμφωνούμε οι δυο μας. Υπενθυμίζω το πλαίσιο σύντομα. Μετά την έγκριση καθυστερημένα <coughs> του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου και των νομικών πράξεων που συνδέονται, πολλά προγράμματα δεν μπόρεσαν να εγκριθούν ε, το 2014 και δεν ήταν αρκετά προηγμένα για να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν με τη μεταφορά πιστώσεων που προβλέπει το άρθρο 13 του Δημοσιονομικού Κανονισμού. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη να τροποποιηθεί το ανώτατο όριο των υποχρεώσεων αν δεν θέλουμε να χαθούν αυτές οι πιστώσεις. Με βάση το άρθρο 19 του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου, τους ώστε αυτές οι χρηματοδοτήσεις που δεν εκταμιεύθηκαν το 2014 να μεταφερθούν στα επόμενα χρόνια. Υπάρχει λοιπόν μια μικρή διάκριση μεταξύ των ε, πιστώσεων που μεταφέρονται με το άρθρο 13 ή της τροποποίησης, όπου δεν χρειάζεται τροποποίηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και διότι αυτές οι πιστώσεις ε, υποχρεώσεων μπορούν να ληφθούν από το 15 λόγω της ευελιξίας που προβλέπει ο δημοσιονομικός κανονισμός και των πιστώσεων που πρέπει να μεταφερθούν επειδή δεν έχει προχωρήσει αρκετά η διαδικασία τους από πλευρά των προγραμμάτων και εδώ υπάρχει υποχρέωση να ζητήσουμε τροποποίηση του πλαισίου, του δημοσιονομικού πλαισίου του πολιτού. Είναι τεχνική φύσης. Δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο ε, μετά τις εκλογές ή ε, κατά το ίμιση της εκτέλεσής του. Αυτή λοιπόν ε, η τροποποίηση αφορά το ΦΕΔΕΡ, το Περιφερειακό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, ε, το Ταμείο Μετανάστευσης, το Ταμείο Ιστορικής Ασφάλειας, την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων. Όλα αυτά τα ταμεία λοιπόν θα τροποποιηθούν και όλα τα κράτη-μέλη. Όλα απαρεγκλήτως στα κράτη-μέλη. Και ως ποσό είναι περίπου το 50% της χρηματοδότησης των ταμείων. Πολύ σημαντικό ποσό δηλαδή. Και κάτι άλλο. Από την τελευταία φορά που το συζητήσαμε, το Συμβούλιο κατέληξε σε άποψη Υπενθυμίζω ότι και στο Συμβούλιο χρειάζεται ομοφωνία για να γίνει αυτή η αναθεώρηση. Στο ΕΚΟΦΗΝ 17 Φεβρουαρίου δόθηκε επί της αρχής συμφωνία για την πρόταση αναθεώρησης και είχαμε δύο δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μία δήλωση πέντε κρατών μελών που συνοδεύουν την απόφαση του Συμβουλίου. Η δήλωση θα σας ενδιαφέρει κύριε Πρόεδρε. Η δήλωση λοιπόν της Επιτροπής προτείνει να χρησιμοποιηθούν όλες οι δυνατότητες ευελιξίας, ιδιαίτερα το συνολικό περιθώριο για τις πληρωμές, που επιτρέπει την υιοθέτηση όλων των μη χρησιμοποιηθέντων περιθωρίων μεταξύ 14 και 15 μέχρι το ανώτατο όριο και η δήλωση της Επιτροπής τονίζει ότι πρέπει να επικυρωθούν τα υπόλοιπα προγράμματα πριν το τέλος του χρόνου για να μην παρεκκλίνουμε από τον προγραμματισμο 14,20. Πέντε μέλη, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία και άλλο ένα, η Ρουμανία, εξέφρασαν κάποιες αμφιβολίες για το εάν και κατά πόσο θα είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν τα επόμενα χρόνια τα ποσά αυτά και ζητούν η Επιτροπή να επιτρέψει μέσω του μηχανισμού αυτόματης ε, εκταμίευσης να ολοκληρωθούν τα προγράμματα. Θα μπορούσαμε να έχουμε πάει πιο γρήγορα, αλλά επειδή θέλαμε να ακούσουμε και την άποψη της ε, Περιφερειακής Επιτροπής, διατηρούμε το χρονοδιάγραμμα ψηφοφοριών της Επιτροπής μας, εάν βεβαίως συμφωνείτε ως σύνολο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Τωμάου. Διευκρινίζω, λέει ο Πρόεδρος, ότι 11 Μαρτίου είναι η προθεσμία υποβολή τροπολογιών, αλλά καταρχήν δεν πρέπει να υπάρξουν τροπολογίε. Την 1η Απριλίου θα ψηφίσουμε για τι ενδεχόμενε τροπολογίε και στην Ολομέλεια θα μπορούσαμε λοιπόν να συζητηθεί σε μήνυ Ολομέλεια για να κερδίσουμε χρόνο. Θέλει κανείς το λόγο από αυτόν. Κανείς. Ωραία, να περάσουμε στο 5. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Χρήστο για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα, την, ε, το Ταμείο για την ε, Παγκοσμιοποίηση. Πρόταση που νομίζω πρέπει να υποστηρίξουμε τη της ελληνικής κυβέρνησης και, της, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Un instant, Monsieur Christos. Vous avez la parole, Monsieur. Vielen Dank. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχα ζητήσει το λόγο, αλλά δεν με είδατε μάλλον. Θα ήθελα για την έκθεση που μόλις ακούσαμε και ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν πολύ αναλυτική, αλλά παρόλα αυτά έχω μία ερώτηση. Σε σχέση με τις μεταφορές πιστώσεων, δεν θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη ότι πριν από λίγο συζητήσαμε αναλυτικά ότι έχουμε πολλούς ε, απλήρωτους ε, λογαριασμούς, τα λεγόμενα resta liquide, RAL, και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι κάνουμε μεταφορές ε, πιστώσεων, πιστώσεων υποχρεώσεων, σαν να μην τρέχει τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα στα τέλη του χρόνου, ότι θα αυξηθούν ακόμη τα ποσά προς ακαθάριση, τα ραλ. Δεν νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε σαν να μην τρέχει τίποτα και να πούμε ότι είναι τεχνική διαδικασία θα πρέπει να σκεφτούμε τι επιπτώσεις έχει αυτό που αποφασίζουμε για τα απλήρωτα κόμποσα, τα ραλ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Αλλά έχουμε μια ομάδα εργασίας ακριβώς για τις πληρωμές. Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εκαθαρίσουμε αυτά τα απλήρωτα ποσά. Να δούμε δηλαδή σε τι στάδιο ε, είναι οι διαδικασίες. Η κυρία Τομά. Ναι, αλλά μία απάντηση, όχι πραγματικά βέβαια απάντηση, αλλά για να αντιδράσω σε αυτό που υπόθηκε. Μα το συμμερίζομαι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ στιγμή δεν προβλέπει μεταφορά πιστώσεων πληρωμών, γιατί δεν ξέρει ακόμη απριόρι το ρυθμό εφαρμογής. Δεν είναι προκαθορισμένος ο ρυθμός πληρωμής αυτών των υποχρεώσεων, αλλά αυτό που θέλω να πω για αυτά που είπατε, όντως για φέτος και για τα δύο-τρία επόμενα χρόνια νομίζω ότι θα μειωθούν οι απλήρωτες, ε, τα απλήρωτα ποσά. Αλλά, αντίστροφα, μπορεί να υπάρξει κατόπιν κατά το 17-18 μία αύξηση, συσσόρευση ακόμη μεγαλύτερη των ποσών προς εκαθάριση. Πρόεδρος, ο καλύτερος τρόπος να μειωθεί η διαφορά μεταξύ υποχρεώσεων και πληρωμών είναι να μεταθέσουμε τις υποχρεώσεις. Αυτό κάναμε το 2014. Γιατί 21 δις δεν δεσμεύτηκαν. Αυτός λοιπόν είναι καλός τρόπος για να μειωθεί αυτή η διαφορά υποχρεώσεων και πληρωμών. Και να διευκολυθούν λοιπόν οι πληρωμές. Αλλά επειδή οι υποχρεώσεις υπάρχουν ακόμη, σε τελευταία ανάλυση κάποια στιγμή θα φράξει το σύστημα. Άρα το πρόβλημα είναι ακόμη μπροστά μας πρέπει να έχουμε μια πολύ καλή εκτίμηση του πώς θα γίνονται οι ροές εκταμιεύσεων. Ξέρουμε τώρα για την πρωτοβουλία των νέων, για παράδειγμα. Το Συμβούλιο αποφάσισε να επιταχύνει τη διαδικασία. Άρα ίσως θα χρειαστούμε περισσότερες χρηματοδοτήσει απλά και μόνο. Λοιπόν, από πλευράς πολιτικού μηνύματο και ο διορθωτικό 1, DAB 1, όχι DAB 2, στον DAB2, τον διορθωτικό προπολογισμό, το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού 2, θα έχετε κάθε δυνατότητα να αποστείλετε και πολιτικά μηνύματα. Ο κύριο Χρήστο έχει το λόγο. Είναι μια πρόταση τη ελληνική κυβέρνηση και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που νομίζω πρέπει να την υποστηρίξουμε ε, και θα σας πω γιατί στην Ελλάδα έχουμε μια μεγάλη κρίση η οποία έχει χτυπήσει φυσικά και την κατανάλωση αλλά και τη διαφήμιση. Και μιλάμε τώρα για 928 άτομα, τα οποία προέρχονται από 16 ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης στην περιοχή της Αττικής, δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά, ε, που χάσαν τη δουλειά τους. Να σας δώσω μερικά στοιχεία για την κρίση στην Ελλάδα. Η διαφημιστική δαπάνη βρίσκεται σήμερα γύρω στο 30% του, του, επίπεδου του 2007. Δηλαδή μέχρι τότε είχαμε μια αύξηση στην κατανάλωση και στη διαφήμιση. Ήταν βέβαια και ένα λάθος γιατί στηρίξαμε την οικονομική ανάπτυξη στην κατανάλωση. Από τότε γίνεται μια φοβερή προσαρμογή η οποία φέρνει αποτελέσματα. Ε, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2009 ήταν 15% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Η Ελλάδα δηλαδή δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της και δανειζότανε και το 2014 έκλεισε με πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 0,9%. Δηλαδή προσαρμοζόμαστε, θα έλεγα, με έναν ε, βίαιο τρόπο στις ανάγκες του διεθνούς ανταγωνισμού και της παγκοσμιοποίησης. Εν πάση περιπτώσει είναι 928 υπάλληλοι, τεχνικοί, δημοσιογράφοι, ε, ραδιοτηλεοπτικών μέσων στην περιοχή της Αττικής που έχουν χάσει τη δουλειά τους και νομίζω πρέπει να τους υποστηρίξουμε. Είναι μια δαπάνη που ξεπερνάει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Θα τους υποστηρίξουμε ε, για να, να προσπαθήσουν να κάνουν ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα το οποίο βέβαια είναι δύσκολο στις σημερινές συνθήκες. Ε, εμείς θα καλύψουμε το 60% των δαπανών και το υπόλοιπο θα το καλύψει ε, το ελληνικό δημόσιο. Ε, νομίζω λοιπόν ότι ε, στα πλαίσια της αντιμετώπισης των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης αλλά και της ενθάρρυνσης της προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας πρέπει να υποστηρίξουμε την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Κίρτσο. Προβλέπετε ανταλλαγή απόψεων. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο παρακαλώ. Ουδής. Το λόγο τότε έχει ο κύριος Χριστοφόρου και πάλι για περίπτωση κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση στην περιφέρεια της Αττικής. Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και αφορά υλοποίηση του αιτήματο της Ελλάδας για χρηματοδότηση συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για 705 απολυθέντες εργαζόμενους στις εκδοτικές δραστηριότητες της περιφέρειας Αττικής. Ύστερα από την εξέταση της αίτησης αυτής, από την Επιτροπή επισημάθηκε ότι ικανοποιούνται πλήρω όλοι οι όροι για να μπορέσει να εφαρμοστούν οι διατάξει και οι κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή. Δηλαδή, ουσιαστικά η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι πληρούνται πλήρω οι όροι που αφορούν για την κάλυψη όλων αυτών των 705 απολυμμένων εργαζομένων που προέρχονται από 46 επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται στον κλάδο εκδοτικέ δραστηριότητε με συνολικό προπολογισμό 6.244.500 εκ των οποίων το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίηση θα συνεισφέρει μόνο το 60%, το άλλο θα το συνεισφέρει το ελληνικό κράτο, δηλαδή 3.776.700. Ο στόχο είναι να μπορέσουν να επαναδραστηριοποιηθούν και να επανενταχθούν στην αγορά εργασία σε αυτέ τι δύσκολε συνθήκε όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι από τον εκδοτικό τομέα. Θεωρούμε ότι η στήριξη αυτού του αιτήματο προέρχεται μέσα από τη συνάφεια των απολύσεων εξαιτία τη παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Και αυτό το γεγονό προκύπτει γιατί στην Ελλάδα από το 2008 υπάρχει μια βαθιά ύφεση με τεράστια ψηλά ποσοστά ανεργία που ξεπερνούν το 30% και με 30% ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται κάτω από το όριο τη φτώχεια. Από το 2008 επιβλήθηκαν τέτοια μέτρα που περιορίστηκε και η ιδιωτική κατανάλωση σε βαθμό που οι πολίτες πλέον ουσιαστικά δεν ε, μπορούν να ανταποκριθούν στα βασικά αγαθά με αποτέλεσμα άμεσα να επέρθει ουσιαστικά σχεδόν χρεοκοπία εις των κλάδων των εκδοτικών επιχειρήσεων σε βαθμό μάλιστα που μέχρι και 60% απόλεσαν τα εισοδήματά τους. Και δεν απόλεσαν μόνο τα εισοδήματά τους αυτός ο κλάδος μόνο από τη μείωση των πωλήσεων αλλά από τα εισοδήματά του και από τη μείωση τη διαφήμιση και από όλε τι άλλε συνέπειε που προήρθαν εξαιτία τη οικονομική κρίση που βαραίνει αυτή τη στιγμή την Ελλάδα. Ένα τελευταίο θέλω να πω γιατί ουσιαστικά με κάλυψε και ο κύριο Κίτσο σε αυτά τα οποία ανέφερε γιατί είναι συναφή, είναι ότι εξετάστηκε πλήρω ότι οι δεσμεύσει του κράτου μέλου τη Ελλάδο θα υλοποιηθούν με τα βεβαιότητος και όσον αφορά την τήρηση των αρχών τη ίση μεταχείριση και τη απαγόρευση των διακρίσεων και όσον αφορά στη συμμόρφωση τη απαιτή που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία και στην νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ότι να μην ληφθεί καμία χρηματοδοτική ενίσχυση από άλλα ταμεία τη Ένωση ή χρηματοδοτικά μέσα, με αποτέλεσμα ουσιαστικά η Επιτροπή, αφού εξέτασε ενδελεχώ όλο αυτό το αίτημα, κατέληξε ότι πληρούνται όλε οι προποθέσει και ότι το αίτημα τη Ελλάδο είναι απόλυτο συμβατό και οφείλουμε να το ικανοποιήσουμε. Πιστεύω είναι δίκαιο αυτό το αίτημα και οφείλουμε να το στηρίξουμε για όλους τους λόγους τους οποίους προανέφερα. Σας ευχαριστούμε. Επιθυμεί να πάρει κάποιο το λόγο για την έκθεση του κυρίου Χριστοφόρου. Αν όχι, περνάμε στην επόμενη έκθεση κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση για την εταιρεία Lufthansa Technique. Το λόγο έχει ο κύριο Νεγκρέσκου. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι Ιρλανδικές αρχές κατέθεσαν ένα αίτημα για τη Lufthansa Technik το Σεπτέμβριο του 2014. Ξεπερνούμε τα 4 εκατομμύρια 2.500 ευρώ, μάλλον 2,5 εκατομμύρια, είναι η ε, συμμετοχή από το ίδιο το Ταμείο. Αναφερόμαστε σε 250 εργαζόμενους εταιρείας αυτής που θα μπορούσαν να υποστηριχθούν με διάφορες υπηρεσίες μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ο αριθμός των πολυμένων εργαζομένων δεν ξεπερνά τον αριθμό των 500 εργαζομένων που προβλέπεται στο Ταμείο. Παρόλα αυτά, η Ιρλανδία μας λέει ότι υφίστανται αυτή τη στιγμή εξαιρετικές περιστάσεις και ότι οι απολύσει αυτέ επηρεάζουν πολύ αρνητικά την τοπική αγορά απασχόληση καθώ επίση και γενικότερα την τοπική οικονομία. Οι Ιρλανδικέ λοιπόν αρχέ ήδη έχουν αρχίσει να παρέχουν υπηρεσίε προ τα άτομα αυτά τα οποία απολύθηκαν ή για τα οποία έπαυσε η σύμβασή τους ή που πρόκειται να πάυσει η σύμβασή του. Θεωρείται λοιπόν ότι πληρούνται οι συνθήκες προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να έχουν ε, πρόσβαση στη χρηματοδότηση που προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμοποίηση. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε λοιπόν όλες αυτές τις πρωτοβουλίες προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να καταφέρουν να ταχθούν εκ νέου στην αγορά εργασίας. Ας μην ξεχνάμε τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται τα άτομα αυτά, συντήρηση για τα αεροσκάφη, ένας τομέας ο οποίος όπως ξέρετε μετεγκαθίσταται όλο και περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τρίτες χώρες. Μέχρι τις 15 Μαρτίου μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες, ενώ ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 23 Μαρτίου στην Επιτροπή Προπολογιστών. Σας ευχαριστούμε. Επιθυμεί να πάρει κάποιος το λόγο. Ο κύριος Δεπρέ, παρακαλώ. Μία ερώτηση ενημερωτική κύριε Πρόεδρε αν κατάλαβα καλά το όσο είπε ο κύριος Νεγκρέσκου, προβλέπεται εδώ πέρα παρέκκληση, καθότι δεν έχουμε φτάσει στον αριθμό των 500 εργαζομένων. Κανονικά για να κινητοποιηθεί το Ταμείο χρειάζονται πάνω από 500 απολύσει. Οι παρεκκλήσεις αυτές είναι συνήθεις, είναι πρώτη φορά προβλέπεται με τέτοια παρέκκληση από τον κανονισμό. Μία ερώτηση αυτή τη στιγμή υποβάλλω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να μας ενημερώσει αν και σε άλλες περιπτώσεις έχει παραχωρήσει μια τέτοια παρέκκληση από τον κανονισμό. Είναι η πρώτη φορά που προβλέπετε κάτι τέτοιο. Πρόεδρος, θα μπορούσε ενδεχομένω να απαντήσει στην ερώτηση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Παραντή ενδεχομένω. Ναι, πρόκειται για πρώτη φορά φέτος. Είναι όντω σπάνιο, αλλά όντω και στο παρελθόν, τα παρελθόντα έτη είχαμε τήσει παρέκκληση. Έχετε λοιπόν την απάντησή σα, λέει ο Πρόεδρος. Παρ' όλα αυτά τίθεται όντω το ζήτημα. Για ποιο λόγο να τίθεται το όριο αυτό των 500 απολυμένων. Ο κύριος Νεγκρέσκου θα λέμε στην έκθεση αυτή ότι δεν θα πρέπει να προκύπτουν συχνά τέτοιε περιπτώσει και θα προτείνουμε επίση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τη το ότι ε, θα πρέπει όντω να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι και αυστηροί κανόνε ώστε να προβλέπεται εφαρμογή τη κινητοποίηση του Ταμείου κατά παρέκκληση. Άλλε ερωτήσει, ε, όχι. Περνάμε λοιπόν στις ψηφοφορίες. Οι ψηφοφορίες όσον αφορά τις μεταφορές πιστώσεων θα γίνουν ηλεκτρονικά. Επομένως να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες σας και να τις αφήσετε στη συσκευή μέχρι το τέλος της διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Παρακαλώ, ε, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Μπορούμε να περιμένουμε μέχρι τις 10.30 ε, για να ξεκινήσει η ψηφοφορία. Αυτό είχε προβλεφθεί άλλωστε αρχικά και κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουν να φτάσουν και οι συνάδελφοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή συμμετέχουν σε εργασίες άλλων επιτροπών. Πρόεδρος, μπορούμε να περιμένουμε. Άλλωστε είναι 10 και 28 και 29, άρα μπορούμε να περιμένουμε μέχρι τις 10.30. Θα ψηφίσουμε καταρχάς ε, για τους προσαντολισμούς τμήμα 3 προπολογισμός 2016. Η συγκητής είναι ο κύριος ε, Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντες. Euh, euh, Θα μπορούσατε κύριε Φερνάντες ενδεχομένως μέχρι τις 10.30 να μας αναφέρετε τις βασικές αρχές που διέπουν την έκθεσή σας. και έχετε δύο λεπτά ακριβώς στη διαθεσή σας κύριε Φερνάντες. Τέσσερα λεπτά, λάθος. Κύριε Fernandez, vous σας έδωσα το λόγο. Ενδεχομένω να μα μιλήσετε λίγα λεπτά πρωτού ξεκινήσει η ψηφοφορία για το περιεχόμενο τη έκθεσή σα. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλες τις ομάδες για τις τροπολογίες που υπέβαλαν και για τη συνεργασία. Και... Πράγματι, αυτή η έκθεση βγήκε ωφελημένη από την συνεργασία όλων. Εγώ είχα ε, δεσμευθεί χωρίς να αλλάξουμε την δομή της έκθεσης, να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον μια καλύτερη ε, συνένεση. Γι' αυτό το λόγο ευχαριστώ πολύ μια ακόμα φορά τους και οδηγητές ε, που εργάστηκαν προκειμένου αυτές οι κατευθυντήριες ε, γραμμές να φτάσουν στην ε, μορφή που έχουν ε, λάβει. Ευχαριστώ πολύ για την ευελιξία που έδειξαν και που χρειάζεται πάντοτε για να βρούμε ένα συμβιβασμό. Σε ένα συμβιβασμό κανείς δεν κερδίζει όλα όσα διεκδικεί. Ελπίζω τέτοιοι, συμβιβασμοί, τέτοιες συνενέσεις να ε, εισακούονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για να χρησιμοποιεί ε, τις προτεραιότητές μας, να λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες μας. Η παρουσίαση αυτού του προσχεδίου τον, από τον Μάιο ε, ήταν χρήσιμη και πιστεύω ότι μας ε, βοήθησε να προχωρήσουμε και να εξελίξουμε ε, τις προτάσεις. Χρειάζεται, λέμε στην έκθεση, να ε, υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν έτσι ώστε το 2016 όλα τα προγράμματα να ε, προχωρήσουν ε, γρήγορα και η εκτέλεσή τους να φτάσει στο σημείο στο οποίο προβλεπόταν ήδη εξ αρχής από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το Συμβούλιο στις δηλώσεις του συνηθίζει να ε, υποστηρίζει την ε, απασχόληση και την ανάπτυξη και ελπίζουμε ότι θα ε, προβλέψει ε, την κατάλληλη χρηματοδότηση έτσι ώστε να γίνει δυνατή η υλοποίηση των υποχρεώσεων οι οποίες έχουν αναλυφθεί. Ελπίζω λοιπόν και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει κάτι τέτοιο Ελπίζω ότι και το σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα υποστηρίξει αυτές τις κατευθύνσεις, ε, έτσι ώστε να κάνει ένα βήμα μπρος όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για να δώσουμε στους πολίτες αυτό που ζητούν επενδύσεις, ανάπτυξη, απασχόληση. Η απασχόληση ιδιαιτέρως ε, αλλά και οι επιχειρήσεις και η επιχειρηματικότητα που πρέπει να είναι πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστώ κύριε Γενική Είναι 10 και 30. Να αρχίσουμε τις ψηφοφορίες. Κάποιος λέει δεν έχει την κάρτα του. Ωραία λέει ο πρόεδρος θα, θα προσμετρήσουμε την ψήφο σας. Ωραία. Κατευθύνες γραμμές για το προπολογισμό του 2016, τμήμα 3. Τροπολογίες 16 και 17 έχουν αποσυρθεί. Τροπολογία 18. Ε, γίνεται πρόταση προφορικής τροπολόγησής της για να προσθέσουμε τις επόμενες λέξεις για ευφυείς, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς προσπάθειες ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει. Ποιοι είναι υπέρ σε αυτή την τροπολογία, αυτή τη τροπολογία 18. Σε ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Α. Εισηγητής υπέρ. Ποια άλλη υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά. Δείς. Αποχές όχι επίσης. Α, δύο αποχές. Εγκρίνεται η συμβαστική α. Στην παράγραφο 1α, τροπολογία 26. Ο συγκητή είναι κατά. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Ευχαριστώ αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 27. Ο είναι κατά. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28. Ο συγητής κατά υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική Β στην παράγραφο 2. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική Β. Τροπολογία 35. Στην παράγραφο 2α. Ο εισηγητής είναι κατά υπέρ. Θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 14 υπέρ 17 κατά μία αποχή. Συμβαστική σε. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Αφορά την παράγραφο 3. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Εγκρίνεται. Στην παράγραφο 3α. Νέα τροπολογία 41. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική D. Στην παράγραφο 4. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά Ευχαριστώ. αποχέ. Η συμβαστική D για την παράγραφο 4 εγκρίνεται. παράγραφο 5. Τροπολογία 50. Συγχτή κατά υπέρ. Θα πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται. Λίγη. Απορρίπτεται. Παράγραφος 5. Τροπολογία 51. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 52. Υπέρ. Υπέρ και ο εισηγητής. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 53 με προφορική τροπολόγηση του εισηγητή. Για το σημείο 6b υπενθυμίζει ότι οι φοροαπάτες και η φοροδιαφυγή επιδρούν αρνητικά στα κράτη-μέλη και την οικονομία τους και κατά συνέπεια και τον προϋπολογισμό. Τονίζει μεταξύ άλλων ότι οποιαδήποτε απάτη του ΦΠΑ όπως ο φόρος του γαϊτανακίου αμέσως επηρεάζει το εισόδημα της Ένωση. Καλεί την Επιτροπή να τονίσει τα κοινοτικά προγράμματα που συμπληρώνουν τη δράση των κρατών μελών στον τομέα. Ο συγκριτή είναι υπέρ, ποια άλλη είναι υπέρ. Ευχαριστώ απόχέ Αποχές. Εγκρίνεται. Περίγραφος 5α, τροπολογία, 54, ε, Συγκριτή κατά υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 5α, τροπολογία 55. Ο συγητής κατά, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στην παράγραφο 6, συμβαστική ε. Υπέρ ο συγητής. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Ευχαριστώ, αποχές. Η συμβαστική ε εγκρίνεται. Στην παράγραφο 6α νέα, συμβαστική F, εισηγητής υπέρ. Άλλη υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Η συμβαστική F εγκρίνεται. Στην παράγραφο 7, συμβαστική G, εισηγητής υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Η συμβαστική G εγκρίνεται. Στην ε, Παράγραφο 7α. Τροπολογία 72. Κατά ο εισηγητή. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Στην παράγραφο 7α. Τροπολογία 74. Κατά ο εισηγητη υπερ Υπέρ παρακαλώ. Άποχε. Άποχες. Απορρίπτεται. Παράγραφος 7α. Αποσύρεται η 75. Παράγραφος 7α. Νέα. Τροπολογία 76. Κατά ο Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 8. Συμβαστική H. Υπέρ ο Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ κατά. Αποχές. Η συμβαστική H εγκρίνεται. Παράγραφος 8α, τροπολογία 85, κατά ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στην παράγραφο 9, συμβαστική I, υπέρ ο εισηγητής, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10, τροπολογία 96 λέει ο Πρόεδρος, ε, υπέρ Ευχαριστώ, κατά, αποχές. 93 λέει τώρα ο Πρόεδρος. Είναι η τροπολογία 93. Τι είπα, λέει ο Πρόεδρος. Τροπολογία 93 εγκρίνεται. Παράγραφος 11. Συμβαστική J. Υπέρος ηγητής. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 12. Τροπολογία 97. Κατά ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 98. Υπέρ ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 13. Τροπολογία 99. Κατά ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 100. Υπέρ ο Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 101. Υπέρ ο Υπέρ. Κατά. <clears throat> Αποχές. Εγκρίνεται. Στην παράγραφο 13α νέα συμβαστική κάπα υπέρωση της υπέρ. Κατά Αποχές. Η συμβαστική ΚΑΠΑ εγκρίνεται. Στην παράγραφο 14, τροπολογία 103. Κατά ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 104. Κατά ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 105. Υπέρ ο εισηγητής. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται 106 κατά ο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται στην παραγοντα 14 14α τροπολογία 107 υπέρ ο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται στην παράγραφο 14α Α, όχι, όχι, όχι. Καλύπτεται. Καλύπτεται από συμβαστικές. Και 108 και 109. Παράγραφος. Περνάμε στην παράγραφο 15, τροπολογία 110. Υπέρ ο εισηγητής, υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται η 110. Περνάμε στην 111. Ο εισηγητής αρνητικός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 112. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 113, παράγραφος 16. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 114, ο εισηγητής είναι κατά. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 115, ο εισηγητής είναι κατά. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Τροπολογία 116 παράγραφος 16α. Υπέρ. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 17 στην, ε, είναι τροπολογία 117. Εδώ λόγο στον εισηγητή για μια προφορική τροπολογία. Ευχαριστώ. Είναι τεχνικής φύσεως να αντικαταστήσουμε post-electoral MFF review, ε, την μετε, ε, τη μετεκλογική εξέταση ε, και, ανα, ε, και τη μετεκλογική αναθεώρηση με το μετεκλογική εξέταση και αναθεώρηση. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 118. Ο εισηγητής είναι κατά. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 119. Ο εισηγητής είναι κατά. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία κατά. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Η ε, ηλεκτρονική επιβεβαίωση για την 120. Scrutin το ouvert. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Παράγραφος 18. Συμβαστική πρόταση L. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος ψηφίζει υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην αιτιολογική έκθεση α, τελική σκέψη α, τροπολογία 1. Ο εισηγητή είναι κατά. Υπέρ, κατά, αποχέ. απορρίπτεται. 2. Ο εισηγητή είναι κατά. Ποιο είναι υπέρ. Κατά, αποχέ. απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ο εισηγητή είναι υπέρ. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη α κεφαλαίο α μικρό. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Η τροπολογία 4 απορρίπτεται. Περνάμε στην ε, τροπολογία 5. Ο εισηγητής είναι κατά. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Ο εισηγητής είναι κατά υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Ο εισηγητής διαφωνεί. ποιο ψηφίζει υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Καλύπτεται από την 7. Η 7 απορρίφθηκε όμως. Περνάμε στην 9. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος ψηφίζει υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Καλύπτεται από τη συμβαστική πρόταση F. Περνάμε στην αιτωλική εκθεση έκθεση C11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 12, ο εισηγητής συνενεί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13, ο εισηγητής συμφωνεί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία... Τροπολογία 14. Ο εισηγητής διαφωνεί Υπέρ. Τροπολογία 14, έτσι. Ο εισηγητής διαφωνεί, λέω. Ποιος είναι υπέρ. Ηλεκτρονική επιβεβαίωση. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 20 υπέρ 13 κατά. Ε, ε, σκέψη D, έκθεση, ε, τροπολογία 15 υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Για το σύνολο του κειμένου, όπως τροποποιήθηκε, ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται το κείμενο 27 ψήφι 5 κατά και μία αποχή. Ο συνάδελφος ο οποίος δεν είχε κάρτα, α, έφυγε. Πήγε να βρει την κάρτα του μάλλον. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Περνάμε στην ψηφοφορία για την ε, κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής και Παγκοσμιοποίησης. Ε, δεν έγινε παρουσίαση των εκθέσεων από τους οπότε καλό τώρα τους ηγητές να πάρουν το λόγο. Ε, έχουμε το Γενικό Γραμματέα στις 11.30, ε, παρακαλώ λοιπόν να είμαστε σύντομοι. Ο λόγος καταρχήν στον κύριο Πλένκοβιτς για την ενό στυλ του Φέρκο NLMK. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Πρόκειται για την πέμπτη έκθεση που αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμής στην Παγκοσμιοποίηση στον τομέα του Χάλιβα και της μεταλλουργίας. Πρόκειται για την περιοχή ενώ ε, εταιρείε ΦΕΡΚΟ και NLMK. Ε, η, κατα... η αίτηση κατατέθηκε από το Βέλγιο το 2013, ακολουθήθηκε η διαδικασία ε, σε συνεργασία μεταξύ Κομισιών και Κοινοβουλίου όλα έγιναν άψογα. Χαιρόμαστε που η διαδικασία που ακολουθείται πλέον είναι πιο γρήγορη. Πρόκειται για ένα ποσό ύψους 981.000 ευρώ Θα είναι σημαντικό το κονδύλιο αυτό για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν από την ανεργία συγκεκριμένων εργαζομένων σε αυτό τον κλάδο στο Βέλγιο. Προτείνω να υποστηρίξουμε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Περνάμε στην ψηφοφορία. Παράγραφος 3, ε, τροπολογία 1, υπέρ ο συγητής. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ο επιχειρησίτης είναι κατά, υπέρ, κατά. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Άρτη ψηφοφορία πέρας. Απορρίπτεται τροπολογία. Τροπολογία 3 με προφορική τροπολογία του εισηγητή, ο οποίος μας προτείνει να αντικαταστήσουμε το κείμενο με το εξή τονίζει την ανάγκη για μια αποτελεσματική και συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να καταπολεμηθεί η ανεργία στον τομέα του Χάλιβα. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται η τροπολογία. Παράγραφος 10α, τροπολογία 4, καλύπτεται όμως. Παράγραφος 12, τροπολογία 5, υπέρ ο υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται η τροπολογία. Παράγραφος 12, α, τροπολογία 6, υπέρ ο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 12β καλύπτεται, η 12γ, τροπολογία 8, υπέρ ο υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 14α, τροπολογία 9, με προφορική τροπολογία του εισηγητή, ο οποίος προσθέτει το εξής, σημειώνει ότι περισσότερο από το ίμιση του συνολικού εκτιμόμενου κόστους θα πρέπει να δαπανηθεί σε υπηρεσίες μετακίνησης, ανάπτυξης και ιδίως σε μέτρα υποστήριξης και επαγγελματικού προσανατολισμού υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Το κείμενο στο σύνολό του όπως τροποποιήθηκε, με ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ, άρτη ψηφοφορία, πέρας. «32 υπέρ, 2 κατά, καμία αποχή εγκρίνεται λοιπόν το κείμενο». Περνάμε για την ψηφοφορία όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, περίπτωση Σαν Κομπάν Securit Βέλγιο. Η κυρία Λιάτ Νιριάντα έχει το λόγο είχα μια τεχνική έκθεση όσον αφορά το EGF, για το οποίο υπήρχε πολύ σημαντική πλειοψηφία και από τα μέλη της ε, Επιτροπής μας. Μειώσαμε λοιπόν το κατόφλι προβλέπεται στους 200 εργαζομένους. Ας μην ξεχνάμε ότι όσοι εργάζονται σε μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν και αυτή πρόσβαση στην απασχόληση, να ξαναβρούν τη δουλειά τους. Θεωρώ λοιπόν θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους 257 εργαζόμενους προβλέπονται στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήθηκε το άρθρο 2 γ καθώς επίσης και τα σχετικά επενδυτικά μέτρα και είναι η τελευταία τέτοια έκθεση η οποία ακολουθεί τον κανονισμό του 2006. Αυτά είχα να πω κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Να, μια δεύτερη εξαίρεση κύριε Παραντή. Σε σχέση με τον κανόνα που προβλέπει κατόφλι 500 απολυμένων. Παράγραφος 1, τροπολογία 3, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 1α, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ, υπέρ ο εισηγητής, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα, κατά ο εισηγητής εδώ, υπέρ παρακαλώ Κατά. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ για αυτό το σημείο. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 17 υπέρ, 13 κατά και 3 αποχές. Παραγράφος 2, τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. αποχές, εγκρίνεται η τροπολογία. Παράγραφος 5, τροπολογία 6, κατά ο εισηγητής, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 6, τροπολογία 7, υπέρ, ο εισηγητής υπέρ παρακαλώ. Κατά. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ναι, είναι τροπολογία 7. Πρόκειται για την τροπολογία παριθμών 7. Συγγνώμη, δεν το ανέφερα, λέει ο πρόεδρο. Παράγραφο 6, τροπολογία 7, υπέρ ο εισηγητή. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρακαλώ. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Η τροπολογία εγκρίνεται. Παραγραφός 6, τροπολογία 8, κατά ο εισηγητής υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10α, τροπολογία 9, υπέρ ο Αποχέ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 11α, τροπολογία 10, υπέρ ο εισηγητης υπερ παρακαλω κατα Αποχέ. υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 12, υπέρ παρακαλώ. Με συγχωρείτε, τροπολογία 11, παράγραφος 12, τροπολογία 11. Πρόκειται για τεχνική διόρθωση η οποία δεν υπόκειται ψηφοφορία. Σας το συγγνωμη συγγνώμη. Παράγραφος 15α, τροπολογία 13, υπέρ ο εισηγητής, υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 17α, τροπολογία 14, υπέρ ο εισηγητής, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1, κατά ο εισηγητής, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ιτολογική σκέψη ε, τροπολογία 2 υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το σύνολο τώρα του κειμένου όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία, άρτη ψηφοφορία, πέρας. Εγκρίνεται το κείμενο 31 υπέρ, 2 κατά, καμία αποχή. Περνάμε στο επόμενο σημείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περίπτωση Αλέο Σολάρη, κυρία Χόφμαν έχει το λόγο. Ναι, πολύ σύντομα η επιχείρηση αυτή έχει έδρα το κράτος του Βρανδεμβούργου και παράγει φωτοβολταϊκά τα οποία όμως δεν μπορούν να ανταγωνιστούν την Κίνα. Η Κίνα παράγει πάρα πολλά τέτοια φωτοβολταϊκά και τα πολύ στην παγκόσμια αγορά. Οι τιμές από το 2010 έως το 2011 έπεσαν κατά 40% το οποίο είναι κάτω από το κόστος ε, πολλών ε, επιχειρήσεων. Ο κύκλος εργασιών συγγνώμη, το κόστος των, ε, της κατασκευής ανέβηκε πάρα πολύ και το τμήμα των φωτοβολταϊκών που παράγει η Γερμανία έπεσε πάρα πολύ. Η Αλέο Σολάρ είναι μόνο μία από τις τέσσερις ε, επιχειρήσεις φωτοβολταϊκών που χρειάστηκε να πτωχεύσουν και να απολυθούν σε Κινέζους επενδυτές. Υπήρξαν γύρω σε 700 απολύσεις και 470 από αυτούς έχουν ήδη μπορέσει να ενταχθούν σε διαδικασίες άλλης απασχόλησης, εξέβρεση άλλης απασχόλησης και σας παρακαλώ να εγκρίνουμε την έκθεση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Βλέπουμε ότι δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το ντάμπινγκ. Άλλο θέμα τώρα είναι αυτό. Παράγραφος 3, τροπολογία 1, υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 έχει αποσυρθεί. Παράγραφος 9, τροπολογία 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 9α, τροπολογία 5, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 10, τροπολογία 6, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 11, αλφα νέα, τροπολογία 7, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 11, β, νέα, τροπολογία 8, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Παράγραφος 11 γάμα νέα. Τροπολογία 9 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 11 δέλτα νέα. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11 ε. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται το σύνολο του κειμένου που τροποποιήθηκε υπέρ, μάλλον ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται το κείμενο όπως τροποποιήθηκε με 30 ψήφους υπέρ και μία κατά. Πάλι κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση για την περίπτωση Σάχεμ Πολωνίας. Σας ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε. Δεν κατεγράφει δική μου ψήφο. Είναι δυνατό να τη συμπεριλάβουμε. Ήμουν κατά. Μπορείτε, παρακαλώ πολύ, να καταχωρήσετε την αρνητική μου ψήφο. Πρόεδρος, πολύ ωραία, τη λαμβάνουμε υπόψη. Ο κύριος Όλμπρικτ κανονικά θα έχει το λόγο για το επόμενο σημείο, αλλά απουσιάζει, άρα μπορούμε να προχωρήσουμε ευθύ αμέσω στην ψηφοφορία. Για την περίπτωση Ιζάχεμ, λοιπόν Πολωνίας, παράγραφος 1, τροπολογία παρεθμών 1, κατά ο εισηγητής υπέρ παρακαλώ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 8, τροπολογία 2, Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα υπέρ είναι Το δεύτερο δε τμήμα καλύπτεται από την παράγραφο 9 και από την προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 8α νέα, τροπολογία 3, υπέρ ο εισηγητής, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 8β νέα τροπολογία 4 υπέρ ο εισηγητής, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Προφορική τροπολογία από τον εισηγητή, ο οποίος μας λέει ότι θα πρέπει να προσθέσουμε στο τέλος της παραγράφου το εξής. Επισημαίνει τη σημασία της διασφάλισης ότι η διπλή χρηματοδότηση σε τέτοιες συμπληρωματικέ δράσεις δεν θα πρέπει να επιτρέπεται. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε, ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται το κείμενο με 29 ψήφους υπέρ, 2 κατά. Μπορέσετε εσείς να ψηφίσετε παρακαλώ. Ωραία. Να περάσουμε τώρα στην ε, περίπτωση Caterpillar. Η κυρία Γέτενμάκη έχει το λόγο. Α, δεν είναι παρούσα. Ωραία, να ψηφίσουμε. Στην παράγραφο 2, α τροπολογία 1, υπέρ, ο υπέρ. Κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 στο παράγραφο 3. Υπέρ ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω. Παράγραφος 4, τροπολογία 3. Ωραία, θα ελέγξουμε, θα ελέγξουμε. Την τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Λοιπόν, με συγχωρείτε. Όντως εγκρίνεται 18-12. Παράγραφος 4, τροπολογία 3, υπέρ ο συγητής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4, τροπολογία 4. Παράγραφος 4α, τροπολογία 4, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5α νέα, τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Τροπολογία 6. Προφορική τροπολόγηση του εισηγητή αντικαθιστά τη λέξη Συμβούλιο με τη λέξη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο εισηγητή ειναι είναι υπέρ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 6α, νέα, τροπολογία 7. Α, καταπίπτει. Παράγραφος 6β, νέα, τροπολογία 8, υπέρ ο εισηγητής, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 7α νέα, τροπολογία 9. Υπέρ ο εισηγητής, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 8, τροπολογία 10. Υπέρ ο εισηγητής, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 9α, τροπολογία 11. Υπέρ ο εισηγητής, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές, Εγκρίνεται. Παράγραφος 9β, τροπολογία 12, υπέρ, ο εισηγητής, υπέρ παρακαλώ. Κατά άποχες. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10, α νέα, τροπολογία 13, υπέρ, ο εισηγητής, υπέρ παρακαλώ. Κατά άποχες. Εγκρίνεται. Το σύνολο του τροποποιηθέντος κειμένου. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται 30 επέρ, 2 αποχές. 2 κατά συγγνώμη 0 αποχές. Και τώρα περίπτωση Αρσελόρ Μιτάλ. Κύριε Νεκρέσκου. Το αίτημα υποβλήθηκε στις 20 Ιουλίου 2014. Σέβεται λοιπόν τους όρους και τις προθεσμίες, συνολικός προϋπολογισμός πάνω από 2,6 εκατομμύρια. 1,5 από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης είναι 1.285 άτομα τα οποία απελήθησαν πάνω από 900 και θα λάβουν βοήθεια μέσω του προγράμματος. Η Επιτροπή και εγώ θεωρούμε ότι αυτή η εφαρμογή σέβεται όλα τα κριτήρια και μπορεί λοιπόν να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση. Παγκοσμιοποίηση. Βάλαμε στην έκθεση το γεγονός ότι η χαλιβουργία έχει πολύ σημαντικά προβλήματα. Πρόσφατα υποβλήθηκαν για τον κλάδο αυτόν τρία αιτήματα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Παρακαλώ για τη στήριξή σας. Πρόεδρος, έχουμε οκτώ τροπολογίες. Όλες ε, είναι υπέροχοι για όλες αυτές. Ε, να τις ψηφίσουμε όλες μαζί για να κερδίσουμε χρόνο. Μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε ήδη επί του συνόλου του κειμένου. Α, πρώτα τι τροπολογίε. Ωραία. Ποιοι είναι υπέρ του συνόλου των τροπολογιών. Ευχαριστώ. Κατά. Όχι, αποχές δεν βλέπω επίση. Ωραία, ενεκρίθησαν οι τροπολογίες. Και τώρα, το, το, το τροποποιηθέν κείμενο, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 29 υπέρ, 2 κατά και 0 απόχες. Ωραία να περάσουμε τώρα στην πρόταση. Τροποποίησης του δημοσιονομικού κανονισμού. Και χαιρετίζω την παρουσία της κυρίας Λαμάρκ που είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Την ευχαριστώ για την παρουσία της. Χαιρετίζω το θεσμικό όργανο και την ε, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα του Ελεκτικού Συνεδρίου. Η κυρία Πρόεδρος Γκρέσλε έχει συντάξει την πρόταση αυτή Μήπως η κυρία Γκρέσλε για να μας παρουσιάσει το κείμενο και τις τροπολογίες. Ε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, ευχαριστώ πολύ όλους τους συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Ερικ Παραντή, ο οποίος ε, συνταξιδοτείται αύριο. Του εύχομαι ό,τι καλύτερο από πλευρά όλων μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Δεύτερον, αφορά την προφορική τροπολογία 6 θέλω να την αποσύρω γιατί έχουν ε, αντιρρήσεις κάποιοι συνάδελφοι είναι στο τέλος τέλος αφορά το άρθρο 196 είναι η τροπολογία 70 είναι προφορική τροπολογία από αυτή της 70 την οποία να αποσύρω ευχαριστώ πολύ μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία ωραία Πάμε. Τροπολογία 30. Ε, ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ. Παρακαλώ σηκώστε το χέρι αν είστε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Ο εισηγητής συμφωνεί. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία Τρία και τέσσερα που είναι ταυτόσιμες για το άρθρο 1 σημείο 1α νέο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφολική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 32 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση α. Ο εισηγητής συμφωνεί υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 και 36. Είναι κοινή ε, ψηφοφορία από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Ο συγητής είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση Β. Ο συγητής συμφωνεί υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. 40 και 41. Ψηφίζονται από κοινού. Πρόκειται για διευκρινήσει, είναι δέσμοι. Ο εισηγητή συμφωνεί υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνονται. Τροπολογία 6. Ο εισηγητή συμφωνεί υπέρ. Κατά. ηλεκτρονική επιβεβαίωση. Άρχεται. εγκρίνεται. Η έξι ήταν αυτή. Περνάμε στην 43. Προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 και 44 είναι ταυτόσιμε ο συγητής συμφωνεί υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνονται. Τροπολογία 8. Ο εισηγητή, όχι, καλύπτεται από τη 44. Τροπολογία 8 και 45 είναι ταυτόσιμες, ο εισηγητής συμφωνεί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 46, ο εισηγητής συμφωνεί, ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 47. Ο συγητής συμφωνεί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το 9, η 9 καταπίπτει. Η 10. Ο συγητής συμφωνεί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 48. Ο συγητής είναι Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 50 και 51 ε, προβλέπεται η προσθήκη της λέξης διαφθορά ε, ως πρόσθετο κριτήριο. Ε, ψηφίζονται ως δέσμοι. Ο εισηγητής συμφωνεί υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 12. Ο εισηγητής συμφωνεί υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση. Ο εισηγητής συμφωνεί. Όχι, συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος, λέει ο Τροπολογία 52. Ο εισηγητή συμφωνεί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Καταπίπτει. 53. Ο εισηγητή συμφωνεί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 54. Ο συμφωνή συμφωνεί. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ε, ναι, ονομαστική ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 13. Ο εισηγητής συμφωνεί. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Ο εισηγητής συμφωνεί υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 καλύπτεται από τη 14. Τροπολογία 15. Ο εισηγητής συμφωνεί υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 καταπίπτει. 16 και 12 είναι ταυτόσιμες. Ο εισηγητής συμφωνεί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 55, ο εισηγητής συμφωνεί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 17, υπέρ ο εισηγητής, υπέρ, Κατά. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Δεκαοκτώ υπέρ 11 κατά μία αποχή εγκρίνεται. Περνάμε στις τροπολογίες 13, 56, 63. Είναι ταυτόσιμες ηγητή συμφωνή. Ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται η 18 καλύπτεται 57 ο εισηγητής συμφωνεί ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 14 ο εισηγητής συμφωνεί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 58 καταπίπτει, η 11 καλύπτεται επίσης, 59 ο εισηγητής συμφωνεί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 61 είναι η προφορική τροπολογία επαρθμών 5 του συντάκτη. Ο εισηγητής συμφωνεί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 64. Ο συμφωνή, συμφωνεί. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Κατά 65. Ο συμφωνή συμφωνεί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 62. Ο συμφωνή, συμφωνεί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 66. Συγείται συμφωνεί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 67. Υπέρ ο εισηγητής. Ποιος ψηφίζει υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Ο εισηγητής συμφωνεί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 68 και 15. Ταυτόσιμες. Ο εισηγητής συμφωνεί. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 69. Καλύπτει από τη 68 και από τη 15. 70, η 70 έχει αποσυρθεί. Όχι. Α, έχουμε, η, η, η προφορική τροπολογία έχει αποσυρθεί. Ψηφίζουμε την 70 χωρίς την τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Έχει καταπέσει. 71 επίση, 72. Και η 16. Είναι ταυτόσιμε. Και θα ψηφιστούν ως δέσμοι μαζί με τις 73, 17, 74 και 18. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος ψηφίζει υπέρ. Κατά. Ε, αποχές. Εγκρίνονται. 75. Καλύπτεται. Τροπολογία 1. Ο εισηγητής συμφωνεί υπέρ κατά αποχές δεν κρίνεται 76 ο εισηγητής συμφωνεί υπέρ κατά αποχές Ωραία, η 19 καταπίπτει, 23 Ο εισηγητής συμφωνεί, υπέρ, κατά, εποχέ εγκρίνεται. Ε, η τροπολογία 25 έχει αποσυρθεί. Περνάμε σε αιτιολογικέ σκέψεις. Τροπολογία 26. Ε, προφορική τροπολογία υπαριθμών 1 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. 19 υπέρ 10 κατά καμία αποχή. Τροπολογία 27, προφορική τροπολογία 2 του εισηγητή, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία αριθμών 1. Καλύπτεται από την 27, 28. Το και οι δύο είναι ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε συμφωνία ο συγητής. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 1 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 και 3 είναι ταυτόσιμες. Συμφωνεί ο εισηγητής υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία. για το σύνολο του κειμένου. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίθηκε με 28 ψήφους υπέρ, μία κατά και μία αποχή. Α, αυτή η ψηφοφορία αφορούσε τις τροπολογίες. Τώρα, η κυρία Γκρέσλερ έχει το λόγο. Yeah, encore ακόμη από αυτού, κύριε Πρόεδρε. Χαίρετε του νομοθετικού ψηφίσματος δηλαδή, με ονομαστική ψηφοφορία. Συγγνώμη, Πρόεδρε, η προηγούμενη ψοφορία που μόλις κάναμε είπατε ότι ήταν για το κείμενο στο σύνολό του. Τώρα όμως μας λέτε ότι αφορούσε τις τροπολογίες. Τι συμβαίνει τελικά. Μιλάμε για την έναρξη διαπραγματεύσεων. Κυρία Γκρέσλε, είναι η εντολή για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Αυτό πρέπει να ψηφίσουμε. Δεν το έχουμε καλύψει αυτό ακόμα. Πρόεδρος, Ξέρετε ότι σύντομα θα ξεκινήσουμε τον τριμερή διάλογο, λέει η κυρία Γκρέσλε. Θα πρέπει προφανώ να έχουμε σύμφωνη γνώμη τη Επιτροπή για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει. Μόλις ψηφίσαμε τις τροπολογίες, και ουσιαστικά κατά αυτόν τον τρόπο δίνουμε επισήμω εντολή για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει. Και ελπίζουμε βέβαια ότι θα ισχύσει η εντολή αυτή. Θα ψηφίσετε διαφορετικά μετά τη διευκρίνηση αυτή, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, ναι, ναι. Αποχή λοιπόν για μένα, Πρόεδρε. Δύο λοιπόν οι αποχές. Πώς είχατε ψηφίσει υπέρ για να αφαιρέσουμε την ψήφο σας αναλόγως. Είχα ψηφίσει κατά, Πρόεδρε, και αυτή τη φορά θέλω να απέχω, εφόσον ψηφίσαμε, όπως είπατε, τις τροπολογίες. Πολύ ωραία. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, ονομαστική ψηφοφορία. Ονομαστική λοιπόν ψηφοφορία, άρθρη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. ...28 πέρα, ένας κατά και μία αποχή... ...και τώρα ψηφίσουμε... ...για την εντολή έναρξης διαπραγματεύσεων... ...με ονομαστική ψηφοφορία, άρτη ψηφοφορία... Πέρας. Εγκρίνεται η εντολή διαπραγματευτική κυρία Γκρέστινε με 27 ψήφους υπέρ και 2 κατά καμία αποχή. Σας ευχαριστούμε πολύ για την εξαιρετική εργασία σας και πραγματικά ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε γρήγορα να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο έχοντας και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού και θέλουμε να μπορέσει να ισχύσει το κείμενο αυτό πολύ γρήγορα και θέλουμε και το Συμβούλιο γρήγορα να καταλήξει σε μια τοποθέτηση για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει. Περιμέναμε πάρα πολύ καιρό ήδη για το κείμενο αυτό. Ενδεχομένω να προβλεφθούν εξαιρετικέ περιστάσει, να χρειαστεί να κάνουμε επιπλέον συνεδριάσει και με την Επιτροπή ΣΕΝΤΕ, ιδίω για ζητήματα εξωτερικών δράσεων. Και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σωστά βέβαια τους δημοσίους πόρους να χαιρετήσω το Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μόλις έφτασε, αλλά έχουμε ακόμα να ψηφίσουμε κάποιες μεταφορές κονδυλίων. Κυρία Γκαρθιαμπάλ Ρουμπιάλα, μπορούμε από εκείνου να ψηφίσουμε όλες αυτές τις αιτήσει μεταφορών. Μπορείτε να μας υπενθυμίσετε λίγο γιατί μιλάμε πολύ γρήγορα. Ναι, είναι πολύ εύκολο. Έχουμε 8 μεταφορές που πρέπει να κάνουμε. Έχουν να κάνουν με το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Δύο από αυτές έχουν να κάνουν με συμφωνίες αλληλείας της Επιτροπής με τη Μαδαγασχάρη και το Πράσινο Ακροτήριο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί όλες. Συμφωνούμε λοιπόν να ψηφίσουμε από κοινού. Καμία παρατήρηση, καμία αντίρρηση. Με ονομαστική ψηφοφορία λοιπόν το σύνολο των ετοιμάτων αυτών μεταφορών. Άρτη ψηφοφορία. Άμα βγάλατε όμως από τη συσκευή την κάρτα σας, σας είχα πει στην αρχή της ψηφοφορίας ότι θα ψηφίζαμε τις μεταφορές με ονομαστική ψηφοφορία και γι' αυτό το λόγο έπρεπε να είχατε αφήσει την κάρτα σας στη συσκευή. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνονται λοιπόν αυτές οι μεταφορές. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Χολμάιερ για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το είχαμε αναβάλει σύντομα γιατί είχα ορισμένες συμπληρωματικές ερωτήσεις. Πρώτον, ε, η μεταφορά για τον διαμεσολαβητή για υπηρεσιακούς λόγους. Μπορεί να υπάρξει ενδεχόμενο να ε, καταργηθεί κάποια ε, θέση και να απολυθεί κάποιος. Υπήρχαν κάποιες τέτοιες ρυθμίσεις. Δεν ήταν θέμα ε, πειθαρχικό ωστόσο, ήταν απλώς υπηρεσιακό, οικονομικά. Βεβαίως αυτό σημαίνει πως θα μειωθούν οι πιστώσεις διότι πρόκειται για την κατάργηση μίας θέσης διευθυντού για υπηρεσιακούς λόγους δεν χρειάζεται λοιπόν να καλυφθεί πλέον η θέση, εφόσον και καταργήθηκε, και θα είναι και πολύ λιγότερες οι μεταβατικές πιστώσεις. Λιγότερες σε σχέση με τον ε, μισθό που είχε προηγουμένως. Άρα δεν έχει καμία αρνητική δημοσιονομική επίπτωση. Οπότε δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω συζήτηση από αυτού. Βεβαίως είμαι υπέρ αυτής της μεταφοράς πιστώσεων και παρακαλώ και την Επιτροπή μας να την εγκρίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, για τις μεταφορές πιστώσεων για τον ευρωπαίδιο Διαμεσολαβητή ψηφίζουμε τώρα με ονομαστική ψηφοφορία, άρτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνονται με 22 ψήφους υπέρ, καμία κατά μία αποχή. Περνάμε στο δικαστήριο αυτή τη στιγμή προκειμένου να δημιουργηθούν αυτές οι νέε θέσει προβλέπουν. Η κυρία έχετε και πάλι το λόγο. Συζήτησα με το δικαστήριο πολύ λεπτομεριακά γιατί για αυτές τις ε, μετακομίσεις θέλουν να κάνουν ε, μεταφορά κάποιων ε, υπηρεσιών του δικαστηρίου που θα ξεκινήσουν το Μάρτιο και το θετικό είναι ότι το Συμβούλιο συμφωνεί με μας ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διότι από το Σεπτέμβριο του 2015 προβλέπονται 12 επιπλέον δικαστές. Οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, οπότε το δικαστήριο θα χρειαστεί να επανέλθει όταν θα έχουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία για τις αναγκαίες πιστώσεις το και το Συμβούλιο επίσης αποφάσισε γιατί δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε 4-5 χρόνια για αποφάσεις του δικαστηρίου, αλλά παρακαλέσαμε το δικαστήριο να υπάρξουν και κάποιες δυνατότητες συνεργασίας να βελτιώσει τη λειτουργία του, ούτω ώστε οι περαιτέρω επιπτώσεις για το προσωπικό από την πρόσληψη νέων ε, δικαστών να μην είναι τόσο υψηλές. Θα επανέλθει λοιπόν ενώπιόν μας ε, το δικαστήριο για να απαντήσει στα αιτήματά μας θα εξετάσουμε τις απαντήσεις, αλλά το κόστος αυτό των μετακομίσεων είναι οπωσδήποτε αιτιολογημένο. Διότι και εμείς είχαμε ζητήσει αυτούς τους νέους, αυτούς τους νέους 12 δικαστές και τον επόμενο χρόνο θα υπάρξουν και άλλοι δικαστές. Γιατί το δικαστήριο ζήτησε επιπλέον θέσεις και συμφώνησε το Συμβούλιο. Συμφώνησε ότι πρέπει να υπάρξει και επαρκής ε, κάλυψη. Χαίρομαι λοιπόν που με την πρωτοβουλία της Επιτροπής Προϋπολογισμών την οποία να ακολουθούμε εδώ και δύο χρόνια και τελευταία είχαμε τονίσει ότι είναι επίγον επιτέλους επιτύχαμε οπότε παρακαλώ την Επιτροπή μας να εγκρίνει και αυτή τη μεταφορά πιστώσεων. Σας ευχαριστούμε κύριε Χολμάιερ. Θα καταφέρουμε λοιπόν να επιλύσουμε το ζήτημα αυτό. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι η Ευρώπη έχει τη γενικότερη τάση να δαπανά δημοσίους πόρους. Χρειαζόταν κανονικά μόνο 12 ή 13 δικαστές, αλλά ήταν αδύνατον για όλο αυτό το χρονικό διάστημα το Συμβούλιο να επιλέξει από ποιε χώρες θα προέρχονταν οι αυτοί 12-13 δικαστές και η λύση ποια ήταν να εγκρίνει 28 επιπλέον δικαστές. Μονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε, άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Ουδής κατά. Εγκρίνονται λοιπόν. Συγχαρητήρια. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την ψηφοφορία. Να καλωσορίσω τον κύριο Κλάους Βέλε, τον Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά από σύσταση του εισηγητή μας, του κύριου Ντεπρέκ, σας καλέσαμε κύριε Γενική Γραμματέα. Δεν ξέρω αν ο κύριος Ντεπρέ θέλει να πάρει το λόγο για κάποιες εισαγωγικέ παρατηρήσεις. Αν όχι, δίνω το λόγο στο Γενικό Γραμματέα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε κύριοι βουλευτές. Μου ζητήθηκε να κάνω μια παρουσίαση για τις κατευθυντήρες γραμμές, δηλαδή οι κύριες κατευθύνσεις, ε, η γενική προσέγγιση, η φιλοσοφία για τον προπολογισμό του 16. Δηλαδή δεν έχουμε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Τα αριθμητικά στοιχεία είναι στην επόμενη φάση εξέταση του προπολογισμού με το οποίο, το προσχέδιο δηλαδή προϋπολογισμού, θα ασχοληθεί το Προεδρείο στις 9 Μαρτίου, μετά θα έχουμε μία συνεννόηση μεταξύ Προεδρείου και Επιτροπής Προϋπολογισμών, τόσο ώστε γύρω στα τέλη Απριλίου, με βάση το αποτέλεσμα αυτής της συνεννόησης, να ε, υποβάλουμε ένα κείμενο στην Ολομέλεια. Φυσικά έχουμε πολύ αναλυτικές συζητήσεις και τον κύριο Ντεπρέ που είναι εισηγητής για τον προπολογισμό. Ήδη από αυτή την ε, πρώτη φάση μερικές ε, εισαγωγικές παρατηρήσεις. Παραδοσιακά, το Κοινοβούλιο λαμβάνει 20% των διοικητικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι μια συμφωνία που ισχύει ήδη 25 χρόνια. Είναι δηλαδή 20% του λεγόμενου κεφαλαίου 5. Οι διοικητικές δαπάνες μπορούν ε, να αυξηθούν με βάση τις δημοσιονομικές προοπτικές της πολιετής με 4,5%. Σημαντικό ποσοστό αν αξιοποιήσουμε πλήρως αυτό το 20%, κάτι το οποίο δεν το κάναμε πέρυσι, θεωρητικά ο προπολογισμό μας θα μπορούσε να αυξηθεί κατά πάνω από 5%. Και η πρόταση που θα κάνω στο Προεδρείο στις 9 Μαρτίου, η πρόταση προπολογισμού που θα κάνω θα είναι για αύξηση γύρω στο 3%. Μπορεί να είναι 2,9, μπορεί να είναι 3,1. Αυτή όμως θα είναι η πρότασή μου στο Προεδρείο αύξηση 3%. Δεν προτείνω λοιπόν να αξιοποιήσουμε πλήρως αυτό το 20% που παραδοσιακά είναι το ποσοστό μας. Για τις δομές τώρα, δηλαδή ποια θα είναι η διάρθρωση των ε, κατευθυντηρίων γραμμών. Αυτό το έχουμε κάνει εδώ και πέντε χρόνια να υποβάλουμε ένα κείμενο τέτοιο. Και επίσης παρουσιάζουμε και τα συγκεκριμένα προγράμματα. Πολλά είναι πολυετή βεβαίως δηλαδή ένα κόστος αφορά ένα κόστος μπορεί να αφορά μια συγκεκριμένη χρονιά, ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό, αλλά είναι πολυετή. Αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο για τα κτίρια. Επίσης, επειδή έχουμε πολλούς νέους βουλευτές, δεν μπορούμε να ξέρουμε εάν όλοι έχουν παρακολουθήσει τις αποφάσεις της τελευταίες πενταετίες. 13 από τους 15 αντιπροέδρους είναι νέοι. Επίσης, στο Προεδρείο και γι' αυτό το σημείωμα που θα υποβληθεί για το θέμα αυτό εξηγεί και πώς έχουμε καταλήξει στην παρούσα κατάσταση. Ποια είναι τα βασικά σημεία. Ένα ιδιαίτερο σημείο, μια ιδιαίτερη προτεραιότητα θα είναι το τομέας της ασφάλειας. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήδη έχουν ε, επέλθει σημαντικές αλλαγές στον τομέα αυτό. Πριν από πέντε χρόνια για την ασφάλεια είχαμε μόνο μία μονάδα, ένα τμήμα, ένα μικρή μονάδα, η οποία μετατράπει σε διεύθυνση, τώρα πλέον σε γενική διεύθυνση. Το προσωπικό αυτής υπηρεσίας σε μεγάλο βαθμό είναι δική μας υπάλληλη διότι στο παρελθόν δεν είχαμε έλεγχο των κεντρικών υπηρεσιών ασφαλείας, διότι ήταν ε, ε, υπεργολαβία αυτό και φέτος θα το κλείσουμε αυτό κυρίως για τις Βρυξέλλες δηλαδή θα επανέλθουν εντός του οργανογράμματός μας οι υπάλληλοι που ασχολούνται με την ασφάλεια δηλαδή οι υπάλληλοι μας γνωρίζουν τους βουλευτές γνωρίζουν το κοινοβούλιο μπορούμε να τους καταρτήσουμε να αισθάνονται ε, πλήρη ότι είναι πλήρως ενταγμένοι στο κοινοβούλιο να μην δουλεύουν δηλαδή εμάς, σε εμά δύο μήνες και μετά δύο μήνες στο Συμβούλιο και μετά στην Επιτροπή, αυτό θεωρώ ότι είναι πραγματική πρόοδος. Παρόλα αυτά, όπως και πριν, υπάρχουν ορισμένες αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και στην κοινή συνεδρίαση που έκανε η δίκηση με τον Προεδρείο τον Οκτώβριο το αναφέραμε. Η μεγαλύτερη αδυναμία είναι η εξωτερική προστασία των κτίριων. Διότι φυσικά ως διοίκηση του Κοινοβουλίου δεν έχουμε την αρμοδιότητα, το δικαίωμα να αναλάβουμε την εξωτερική ασφάλεια. Εδώ χρειαζόμαστε συνεργασία των κρατών που μας φιλοξενούν στο Βέλγιο ή στη Γαλλία. Στη Γαλλία, στο Στρασβούργο είναι αρκετά καλά ανεπτυγμένη η κατάσταση. Στο Βέλγιο όμως μέχρι πριν από λίγο ήταν ιδιαίτερα ανεπαρκής η κατάσταση και μετά τα τελευταία γεγονότα ξέρουμε ότι η προστασία δεν μπορεί να ξεκινάει εντός του κτηρίου. Η προστασία, η ασφάλεια πρέπει να ξεκινάει εκτός του κτηρίου. Εάν ο κίνδυνο ε, ήδη έχει μπει στα κτίρια μα είναι πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση. Γι' αυτό κάνουμε πολύ λεπτομεριακέ συζητήσει με το βαλγικό κράτο, που ήδη έλαβε μερικά πρώτα θετικά μέτρα, ούτω ώστε να βελτιωθεί η εξωτερική προστασία των κτίριων μα. Ιδεοδό, αυτό θα πρέπει να ισχύσει για όλα τα θεσμικά όργανα. Δεν θέλουμε ειδική λύση για το Κοινοβούλιο, πρέπει να ισχύσει και για τα τρία θεσμικά όργανα. Επιτροπή και Συμβούλιο να μην υπάρχει διαφορά στο επίπεδο προστασίας μετά την ε, παρούσα κρίση να μην επανέλθουμε στο προηγούμενο status quo. Αυτός είναι ο στόχος μας. Επιπλέον, πρέπει να εξετάσουμε τις εγκαταστάσεις ασφαλείας ε, στις εισόδους του κτηρίου μας, ιδίως το κτίριο ASP πρέπει να γίνουν πολύ καλύτερες, να βελτιωθούν πολύ. Οι εγκαταστάσεις που έχουμε τώρα δεν είναι η τελευταία λέξη. Θα πρέπει λοιπόν, αν κάποιος καταφέρει ακόμη και να μπει στο κτίριο, να μπορεί να γίνει ουσιώδης έλεγχος, δηλαδή να μην μπορεί μόλις μπει στο κτίριο να μπορεί να μπει στους κεντρικούς χώρους του κτιρίου. Αυτό αποφάσισε το Προεδρείο, το Προεδρείο στην τελευταία του συνεδρίαση. Για παράδειγμα, θα αυξηθούν κατά πολύ τα τζάμια τα οποία χωρίζουν τμήματα του κτιρίου και ε, αυτές ε, οι βιτρίνες θα είναι αλεξίσφαιρες. Όλα αυτά βεβαίως ε, έχουν υψηλό κόστος που θα συμπεριληφθεί στον προπολογισμό του 16. Θα κάνουμε επιπλέον ε, προσπάθειες να εγκαταστήσουμε αυτές τις νέες εγκαταστάσεις όσο δυνατόν ταχύτερα και ορισμένα μέτρα τα οποία προβλέπαμε για το 2015 να τα αναβάλουμε για το 2016. Γιατί τα μέτρα βελτίωση των εγκαταστάσεων ασφαλείας είναι η απόλυτη προτεραιότητα. Επίσης πρέπει να επενδύσουμε στον τομέα της πληροφορικής. Έχουμε 16 διαφορετικά λογισμικά για την ασφάλειά μας, τα οποία δεν επικοινωνούν ε, βελτίστως. Θα πρέπει να αντικατασταθούν με ένα λογισμικό, ένα σύστημα, όπου να εισραίουν όλες οι πληροφορίες. Αυτό σημαίνει δαπάνες. Επίσης, κατά την επόμενη συνεδρίαση του Προεδρείου προβλέπεται, ελπίζω να προλάβουμε το συζητήσουμε αλλιώς στην μεθεπόμενη, είναι το θέμα των καρτών εισόδου, των badge. Ε, είναι πεπαλαιωμένα αυτά τα badge τεχνολογικά, χρειαζόμαστε νέου τύπου, ήδη χρησιμοποιεί νέου τύπου κάρτες Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να καθορίσουμε ποιες πληροφορίες πρέπει να περιέχουν αυτές οι κάρτες, πώς θα έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, αυτά είναι ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία, οπότε πρέπει οπωσδήποτε να τα συζητήσει και το Προεδρείο πριν ληφθεί η τελική απόφαση. Αλλά θεωρώ ότι το Προεδρείο μάλλον στην επόμενη συνεδρίασή του στις 9 Τρίτου θα αποφασίσει αλλιώς τον Απρίλιο. Αυτό θα έχει επιπτώσεις στον προπολογισμό του 16. Το άλλο θέμα που θέλω να αναφέρω είναι το επίδομα γραμματείας. Έχουμε παγώσει τα επιδόματα τα τελευταία χρόνια. Η τελευταία αξιόλογη αύξηση των επιδομάτων γραμματείας έγινε το 10 και το 11. Τότε είχαν αυξηθεί κατά 1500 ευρώ. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι για το επίδομα γραμματείας, αυτό είναι βέβαια μια πολιτική απόφαση, τότε η σωστή χρονιά γι' αυτό θα ήταν το 16. Για το 16 μπορούμε να φέρουμε επιπλέον έξοδα. Δεν χρειάζεται να πληρώσουμε μεταβατικές ε, πληρωμές για τους νέους ε, βουλευτές, λίγοι θα αλλάξουν, ούτε έχουμε τις ιδιαίτερες δαπάνες που έχουμε όταν ε, έχουμε εκστρατείες για ευρωεκλογές είναι μια πολιτική απόφαση, άρα πρέπει να ληφθεί από το Προεδρείο. Το περιθώριο ελιγμό στον προπολογισμό υπάρχει, προβλέπεται. Αλλά πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Προεδρείο. Και κατόπιν ενδεχομένω θα έχει δημοσιονομικέ επιπτώσει. Τρίτον, για τα κτίρια και υπηρεσίε επιμελητία, στήριξη. Από το 19 θα πρέπει να ε, έχουμε ανακαίνιση του κτηρίου Polan ε, Μία εμπειρογνωμοσύνη που είχαμε πρόσφατα μας είπε ότι είναι πήγουσα η ανάγκη ανακαίνισής του, συντήρησής του και αυτά που διαπιστώσαμε με την οροφή του ημικυκλίου στις Βρυξέλλες ε, μας δείχνει ότι πρέπει να γίνουν ε, βελτιώσεις. Και όλο το σύστημα της ίδρευσης και του ηλεκτρισμού, ε, των σωλήνων δηλαδή και των καλωδίων, μας έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα και έχουμε βλάβες συχνά. Βέβαια μπορούμε να κάνουμε ε, επισκευές, αλλά πρέπει οπωσδήποτε πριν την επόμενη κοινοβουλευτική θητεία να έχουμε προβλέψει μία συντήρηση. Οπότε καλό είναι να υπολογίσουμε από το παρελθόν, δηλαδή να έχουμε μία προσέγγιση πολυετή ούτω ώστε να μπορούμε το 19 να ξεκινήσουμε αυτή την ανακαίνιση. Έχουμε 600 γραφεία, έχουμε την αίθουσα της Ολομέλειας, έχουμε άλλες αίθουσες συνεδριάσεων και έχουμε και κοινόχρηστους χώρους για εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα ο χώρος για Χούντι Αυτά τα, αυτές οι εγκαταστάσεις, αυτοί οι χώροι δεν μπορούν να μην λειτουργούν λόγω επισκευών εάν δεν έχουμε εναλλακτικού χώρου για τι εκδηλώσει των βουλευτών. Δηλαδή χρειαζόμαστε ένα σταδιακό σχέδιο για το πώ θα συντηρηθεί κατά τμήματα αυτό το κτίριο. Η ομάδα εργασίας μας για τα κτίρια έχει εκπονήσει μία μεσοπρόθεσμη στρατηγική για τα κτίρια διότι η προηγούμενη μεσοπρόθεσμη στρατηγική μας για τα κτίρια ήταν από το 2010. Τώρα λοιπόν πρέπει να εκπονήσουμε μια στρατηγική για τα κτίρια για αυτήν την παρούσα κοινοβουλευτική θητεία, η οποία να προγραμματίσει τις ανάγκες μας χρόνο το χρόνο, όλα τα μέτρα μας για τα κτίρια, είτε πρόκειται για νέα κτίρια, είτε πρόκειται για συντηρήσεις, είτε πρόκειται για μισθώσεις, έχει μια προκατακτική διαδικασία. Και πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν να ληφθούν οι αναγκαίε αποφάσει. Είχαμε δυνατότητα στην αρχή αυτή τη θητεία να βελτιώσουμε κάπως την κατάσταση για τα γραφεία των βουλευτών και των, συνεργαζών, και των συνεργατών τους. 1.200 ε, ε, πάλι πήγαν στο κτίριο της πλατείας Ντεμέους, κάτι που επέτρεψε να δώσουμε στους βουλευτές 450 επιπλέον γραφεία. Βέβαια η κατάσταση για ορισμένους βουλευτές προηγουμένως ήταν τραγική είχαν 5-6 συνεργάτες σε ένα γραφείο. Αυτό δεν θα το επέτρεπε φυσικά η Βελγική, δεν το επέτρεπε η Βελγική νομοθεσία. Δώσαμε λοιπόν 450 ε, νέα γραφεία σε 450 βουλευτές. Αυτό σημαίνει, άμα κάνεις το λογαριασμό, ότι 300 ε, είναι ακόμη με την προηγούμενη κατάσταση. Είναι λοιπόν αυτό ένα θέμα που πρέπει να το δούμε τα επόμενα χρόνια και να το λύσουμε. Τώρα, γενικά η επίπλωση. Η επίπλωση θα είναι 20 ετών το 16. Σταδιακά λοιπόν και εδώ πρέπει να αντικατασταθεί η επίπλωση, ο εξοπλισμός συνολικότερα. Αυτό πρέπει να γίνει για να επιτρέψει περισσότερη ε, ευελιξία χρήσης των γραφείων. Διότι αυτή τη στιγμή σε κάθε βουλευτή προσφέρουμε ακριβώς τον ίδιο εξοπλισμό, αλλά οι ανάγκες των βουλευτών δεν είναι ίδιες. Είναι ορισμένοι που θέλουν ένα γραφείο για συνεδριάσεις, είναι ορισμένοι που θέλουν να αλλάξουν την κατάσταση, να μπορούν να αλλάζουν την κατάσταση όταν είναι παρόντες και όταν λείπουν. Θέλουμε λοιπόν να είναι πιο ευέλικτη η προσφορά εξοπλισμού. Ούτω ώστε κάθε βουλευτή ανάλογα με τι ανάγκε του να μπορεί να καθορίσει πώς θα διαμορφώσει το γραφείο του στα πλαίσια βέβαια ενός συγκεκριμένου κόστους με κάποιο περιορισμό στις εναλλακτικέ λύσεις αλλά υπάρχουν τώρα νέοι τρόποι επίπλωσης και διαμόρφωση των γραφείων που επιτρέπουν μεγάλη ευελιξία και όταν αντικαταστήσουμε τα έπιπλα τότε πρέπει να το συνδέσουμε με αυτήν την κάποια ευελιξία. Είναι ένα θέμα που το μελετάμε αυτή τη στιγμή αλλά θεωρώ ότι ήδη από το 16 θα παίξει ρόλο στον προπολογισμό. Το προηγούμενο Προεδρείο είχε αποφασίσει μια νέα στρατηγική για τα εστιατόρια, για τις καντίνες. Η κατάσταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ότι έχουμε μόνο έναν ο οποίος έχει όλα τα εστιατόρια μονοπωλιακά. Αυτό δεν είναι ποτέ καλό. Είναι καλύτερο να υπάρχουν διάφοροι, να μπορούμε να επιλέξουμε Γι' αυτό υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί τεχνικοί. Μέχρι στιγμή είχαμε μόνο μία κουζίνα, για παράδειγμα. Ένα μόνο μαγειρίο. Θέλουμε λοιπόν να περάσουμε από την κατάσταση όπου ένας, μία επιχείρηση είχε όλα μας τα εστιατόρια σε μια κατάσταση όπου θα υπάρχουν διάφορες επιχειρήσεις στα εστιατόρια μας. Και μετά να περάσουμε σε μια κατάσταση όπου θα έχουμε πολλές επιχειρήσεις που να έχουν τα εστιατόρια μας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με τη μία, διότι όπως σας είπα έχει να κάνει και με τον εξοπλισμό των μαγειρίων, αλλά οι νέες προκηρύξεις θα γίνουν με τέτοιο τρόπο, ούτω ώστε να μην είναι δυνατόν να έχουμε μονοπωλιακές καταστάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε διάφορες επιχειρήσεις ε, εστίασης με διαφορετικές αντιλήψεις. Και θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα έξοδα. Στον προπολογισμό, ο προπολογισμό να καλύπτει όλα τα έξοδα τη εστίαση. Τώρα, στον τομέα των δημοσίων σχέσεων και της επικοινωνία, Ξέρετε ότι το Μάιο του 2014 για πρώτη φορά είχαμε την ε, εκδήλωση αυτή για την νεότητα με 5-6 νέου από όλε τι χώρε τη Ευρώπη που έλαβαν μέρος και οι αντιδράσεις ε, που είχαμε, ο αντίκτυπος ήταν απόλυτα θετικό και χαίρομαι που ε, τώρα έχουμε νέους που κάλεσαν διάφορους ε, από τους ε, συμμετέχοντες σε αυτή την εκδήλωση για να ακούσουν τις απόψεις τους ε, και τις προτάσεις τους. Και είχε πολύ θετικό αντίκτυπο και αυτή η πρωτοβουλία. Το Προεδρείο λοιπόν αποφάσισε να επαναληφθεί αυτή η εκδήλωση το 2016 στο Στρασβούργο. Πρέπει λοιπόν και αυτό να το συμπεριλάβουμε στον προπολογισμό. Ο οίκος της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, το σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Υποθέτω ότι οι εργασίες διαμόρφωσης του κτηρίου, οι καθαρά οικοδομικές εργασίες ε, θα λήξουν πριν το καλοκαίρι, οπότε το Σεπτέμβριο θα μπορέσουμε να βάλουμε και τις τζαμαρίες γύρω από το κτίριο, αλλά αυτό δεν επηρεάζει τις εργασίες στο εσωτερικό, οπότε μετά θα έχουμε ένα χρόνο για να αποφασίσουμε τις εκθέσεις. Να αποφασίσουμε το περιεχόμενο δηλαδή. Οπότε το καλοκαίρι του 2016 αναμένω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε τα εγγένεια. Στον προπολογισμό λοιπόν του 2016 ε, σημαίνει ότι θα υπάρξουν κάποιες συγκεκριμένες δαπάνες, δεν θα είναι πια οικοδομικές δαπάνες, αλλά ε, για το περιεχόμενο. Τα αντικείμενα, τα εκθέματα. Βέβαια από κάποια εκθέματα, για κάποια εκθέματα είμαστε εμείς ιδιοκτήτες, οπότε δεν θα έχουμε έξοδα. Και το Κοινοβούλιο επίσης, ε, επίσης αποφάσισε να υπάρξει ένα καλύτερο λογότυπο του Κοινοβουλίου που να είναι καλύτερο και για την ηλεκτρονική επικοινωνία. Αυτό το λογότυπο το εκπονήσαμε εμείς οι ίδιοι μαζί με το Γραφείο Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δεν είχε υψηλό κόστος. Αλλά το ενέκριναν παρόλα αυτά τα μέλη του Προεδρείου, παρά το χαμηλό του κόστος, άρα μπορούμε να κάνουμε περισσότερο εμεί ίδια από ό,τι νομίζουμε. Δεν θα μας... Ε, δεν θα επιφέρει η εισαγωγή του έξοδα, δηλαδή θα αξιοποιήσουμε όλα τα έγγραφα, όλους τους φακέλους, ε, όλο το χαρτί με το παρόν λογότυπο μέχρι τέλους και μετά θα εισαγάγουμε το νέο, μόνο για κάποιες εκδηλώσεις θα έχουμε το καινούριο. Το θα έχουμε και το νέο ασφαλέστερο κέντρο για υποδοχή επισκεπτών, διότι η κατάσταση τώρα είναι ότι έρχονται τα πούλμαν με τους επισκέπτες και τους αφήνουν, και τους αφήνουν στη βροχή. Πρέπει να κατέβουν οι επισκέπτες από τη βροχή. Ενώ τώρα θα, τα λεωφορεία θα μπορούν να φτάνουν ακριβώς έξω από το κτίριο και από το Παρλαμεντάριο. Από το 16 λοιπόν θα έχουν λήξει αυτές οι προσαρμογές. Για το 16 επίσης θα έχουμε με τα εγγένεια του σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας ένα πλήρη κύκλο επισκέψεων που θα μπορεί να κάνει κανείς και θα είναι δυνατόν και άτομα με προβλήματα κινητικότητας, ε, ηλικιωμένα άτομα, οικογένειες, όλοι αυτοί θα έχουν άνετη πρόσβαση. Θέλουμε όλοι να επισκέπτονται, ε, να έχουν δυνατότητα να πάνε σε όλα αυτά τα κτίρια. Αυτή τη στιγμή θα διαπιστώσετε ότι όποιος ε, θέλει να πάει στο σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας πρέπει να κατέβει μια πολύ απότομη σκάλα Θέλουμε λοιπόν να λύσουμε τα προβλήματα αυτά, ούτως ώστε να μπορούν όλοι να επισκεφθούν και αυτό τον χώρο. Δεν έχουμε λάβει ακόμη ως Προεδρείο λεπτομερικές αποφάσεις. Τώρα για τις ειδικέ εκθέσεις και μελέτες που ε, παραγγέλνουμε. Πολλές επιτροπές έχουν ήδη πολλούς εμπειρογνώμονες ε, στις γραμματείες τους και έχουμε και την υπηρεσία μελετών, η οποία και εκείνη μπορεί να κάνει εκθέσεις. Αυτό είναι πολύ ουσιώδες για να είμαστε βεβαίως ισότιμα, ισότιμος παράγων στην ε, θεσμική διαδικασία, να μην εξαρτώμεθα μόνο δηλαδή από εξωτερικές υπηρεσίες. Όμως έχουμε κάποια προβλήματα για κάτι συγκεκριμένο. Δεν έχουμε ακόμη επαρκή εμπειρογνωμοσύνη, είναι ο τομέας των κατεξοδότηση πράξεων. Για παράδειγμα, οι οικονομικές επιτροπές μετά τη χιονοστιβάδα νομοθετημάτων των τελευταίων ετών θα λάβουν τώρα γύρω στα 400 κείμενα κατεξοδότηση πράξεων και εφαρμοστικών πράξεων. Είναι νομοθετήματα όμως και αυτά. Το Κοινοβούλιο μπορεί να σχολιάσει και να αρνηθεί. Έχει ευθύνη για αυτά τα κείμενα. Δηλαδή το Κοινοβούλιο όταν ενέκρινε να υπάρξουν εξοδότηση πράξης ενέκρινε επιπλέον αρμοδιότητες για τον εαυτό του. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε εάν και κατά πόσο συμφωνούμε με αυτές τις πράξεις. Αυτό θα είναι μεγάλο πρόβλημα για τις οικονομικές επιτροπές, επειδή όπως είπα είχαμε αυτή τη χιονοστιβάδα νομοθετημάτων, τώρα έχουμε μια δεύτερη χιονοστιβάδα εφαρμοστικών και κατοξιοδότηση πράξεων. Είχαμε παρόμοιο πρόβλημα για τα θέματα περιβάλλοντος όπου υπήρξαν περίπου 600 τέτοιες πράξεις το χρόνο. Τώρα θα έχουμε λίγο λιγότερες λοιπόν, αλλά είναι πολύ σημαντικές αυτές οι πράξεις για τη βιομηχανία, τις μεταφορές. Θα προτείνω λοιπόν στο Προεδρείο να υπάρξουν ε, κάποια μικρά τμήματα όπου να γίνεται κάποια προπαρασκευή για τους βουλευτές για να μπορούν να λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις. να μην αφήνουμε να περνάνε δηλαδή τέτοιε πράξει, δηλαδή να μην αφήνουμε να περνάνε νομοθετήματα χωρί ο νομοθέτη να μπορεί να εξετάσει στην ουσία τα θέματα. Και ξέρω ότι αυτό είναι το αίτημα και του συγκεκριτή κυρίου Ντεπρέ. Κάτι το πρώτελευταίο για τι γλώσσε. Τα τελευταία χρόνια επιτύχαμε πολλέ αυξήσει τη αποδοτικότητά μα και νομίζω ότι μεταξύ των οργάνων είμαστε αυτοί που έχουν την πιο αποδοτική τις πιο αποδοτικές γλωσσικές υπηρεσίες θα πρέπει να κάνουμε περαιτέρω επενδύσεις στην τεχνολογία, για παράδειγμα για τη μετάφραση. Από 13 σελίδες κείμενο που μπορεί να λάβουμε, 5 από τις 13 σελίδες δεν χρειάζεται να μεταφραστούν, αναγνωρίζονται από κάποια λογισμικά επειδή είχαν προκύψει σε άλλα κείμενα και έχουν ήδη μεταφραστεί. Δηλαδή ένα μεγάλο τμήμα της μετάφρασης ε, το κάνει ο υπολογιστής βέβαια μετά πρέπει να ελεγχθεί. Αλλά 5 από τις 13 σελίδες κατά μέσο όρο να μεταφράζονται αυτόματα αυτό σημαίνει εξοικονόμηση ενέργειας και αυτό μπορούμε να το αυξήσουμε εάν κάνουμε τις αναγκαίες επενδύσεις στην σχετική τεχνολογία. Πρέπει να το κάνουμε. Παλιότερα είχαμε 1200 μεταφραστές Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να περιορίσουμε το φόρτο εργασίας και το προσωπικό πρέπει να το χαιρετήσουμε. Επίσης να σας πω ότι ε, γίνονται διαπραγματεύσεις μεταξύ των διερμηνέων μας και της Γενικής Διεύθυνσης για να υπάρξουν ε, πιο ευέλικτες ε, μορφές και πιο ευέλικτα ωράρια εργασίας. Έχουμε μια προσωρινή συμφωνία μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης και των διερμηνέων και αυτή η ευελιξία θα μας βοηθήσει σε περαιτέρω εξοικονομήσεις ούτω ώστε να διατηρήσουμε την πολυγλωσία σε όλες τις γλώσσες και να μπορούμε να τη χρηματοδοτήσουμε. Και κάτι τελευταίο για τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού. Τα επόμενα χρόνια θέλουμε ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών. Δεν έχουν τώρα έτσι τα πράγματα. Μόνο κάποια τμήματα, κάποιες διαδικασίες έχουν προχωρήσει. Άλλοι είναι ακόμη στη δεκαετία του 70 ή του 80 αν θέλω να είμαι γενναιόδωρος. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια συνεπής ψηφιοποίηση, ψηφιακοποίηση και ο νέος γενικός διευθυντής θα το επιχειρήσει, θα πάρουμε κάποια συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν θα έχουμε λοιπόν κόστος ε, εισαγωγής νέου λογισμικού. Παράδειγμα, στον τομέα των βοηθών. Είχαμε 1.709 συμβόλαια το προηγούμενο εξάμεινο και είχαμε βέβαια και τη λήξη συμβολέων άλλων βοηθών. Είναι αυτός ένας τεράστιος όγκος εργασίας, γι' αυτό χρειαζόμαστε σύγχρονη πληροφορική, σύγχρονη μηχανοργάνωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε και Γραμματέα για την παρουσίαση αυτών των ε, κατευθύνων γραμμών του προϋπολογισμού. Ε, η αξιοπιστία μας ε, εξαρτάται από τον καλό χειρισμό των πόρων μας. το Κοινοβούλιο πρέπει να αποτελεί υπόδειγμα διαχείριση. Ε, τον κύριο Βίλαντ που είναι αντιπρόεδρο, υπεύθυνο για τον προπολογισμό. Είχαμε προβλέψει την παρουσία του τον Μάρτιο για την παρουσίαση του ε, προσωρινού προπολογισμού του Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε κύριε Γενική Γραμματέα. Αν μας επιτρέπετε να σας θέσουμε κάποιες ερωτήσεις. Ο λόγος του κύριο Μάνκα.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 Είχατε μεγάλα σχέδια για την, ε, για την ασφάλεια, για την υπηρεσία ασφάλειας από το 2010. Ήδη έχουν γίνει πολλά. Έγινε γενική, γραμμα, γενική διεύθυνση. Ως εισηγητής ε, σας ε, ε, είχα ζητήσει πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, μια, ένα έλεγχο, εσωτερικό έλεγχο στην Γενική Διεύθυνση in Law. Ε, δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά μήπως θα μπορούσατε να μου πείτε ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου που είχαμε ζητήσει. Σήμερα αναφερθήκατε σε μια στρατηγική για το μέλλον. 3% αύξηση προφανώς εξαρτάται από τα διάφορα, από το πρόγραμμα εργασίας μας, από τα διάφορα σχέδια τα οποία να συζητήσουμε. Ε, θα μπορούσα να προτείνω και κάποιες επιπλέον περικοπές και εξοικονομήσεις θυμάστε ότι στο παρελθόν κάναμε διάφορες αξιολογήσεις και είχαμε δει ότι θα ήταν καλύτερο το κοινοβούλιο να κατέχει τα κτίρια και όχι να τα νοικιάζει. Η ανάλυση είχε δείξει ότι από οικονομικής πλευράς ε, είναι καλύτερη η κτίση τους και ε, από την ενοικίασή τους. Δεδομένου ότι έχουμε μόνο μια πηγή κτηρίων. Ε, ο κίνδυνος ήταν ε, οι τιμές να είναι υψηλές. Ε, εσείς είπατε ότι οι πλειώνες προμηθευτές είναι ε, καλό πράγμα γιατί μειώνει τις τιμές. Οπότε θα πρέπει να, το κάνουμε το ίδιο, να κάνουμε το ίδιο πράγμα ακριβώς και στην απόκτηση κτηρίων. 409 βουλευτές ε, συνταξιοδοτήθηκαν ε, αμέσως μετά τις ε, τελευταίες εκλογές γιατί δεν επανεκλέγησαν. Και λέτε ότι από αυτό θα προκύψουν εξοικονομήσεις 1,8 εκατομμύρια ευρώ συγκεκριμένα δεν θα χρειαστούν το 2016. Και αυτό μας δίνει ένα αποθεματικό που μπορεί να δαπανηθεί αλλού. Είχα πει και στο παρελθόν ότι τον Ιανουάριο ε, υπέβαλαν 1.216, 1.563 ε, και 563 αιτήματα. Ερωτήσεις στην Επιτροπή. Ε, με κόστος σχεδόν 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Πόσο από αυτό το κόστος το αναλαμβάνει το Κοινοβούλιο και πόσο η, η Κομισιόν. Μερικές φορές ε, τα μέλη ε, θέτουν ερωτήσεις για να αυξήσουν απλώς ε, το νούμερό τους για να φαίνονται πιο ψηλά στον κατάλογο. Γιατί παίρνουν πόντους για ερωτήσεις που βάλουμε μπλε κάρτα Δεν πρέπει όμως ε, να κάνουμε ερωτήματα μόνο και μόνο για να βελτιώνουμε το προφίλ μας, τα στατιστικά μας. Οι ερωτήσεις, τα ερωτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται ασφαλώς ε, σε επιτρόπους, αλλά αν δεν δημοσιεύονται στο... Αν δεν δημοσιευόντουσαν στο ίντερνετ θα γλιτώναμε ένα μεγάλο ποσό. Πόσο πληρώνεται από την Κομισιόν και πόσο μας κοστίζει εμάς αυτή η διαδικασία, όπως ξέρετε. Είπα επίσης ότι το Κοινοβούλιο είναι υποχρεωμένο να μεταφράζει όλες τις τροπολογίες. Όλες τις τροπολογίες θα πρέπει να μεταφράζονται στις γλώσσες αυτής και των άλλων επιτροπών. Μερικές φορές οι μεταφράσεις δεν γίνονται έγκαιρα. Και μερικές φορές οι τροπολογίες είναι όλες σε μία γλώσσα. Είχαμε ψηφίσει ακόμα και αυτές που απορρίπτονται να μεταφράζονται σε όλες τις γλώσσες. Δεν είναι λογικό αυτό, δεν χρειάζεται, είναι περιττό. Μαζί με τον εισηγητή είπαμε ότι αποδείξαμε ότι θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε εκατομμύρια ευρώ από αυτό το θέμα. Ε, αυτή είναι η τρίτη μου θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ποτέ δεν έχω διαβάσει τα, ε, το τα verbatim πρακτικά των συνεδρίασεων. Δεν ξέρω, υπάρχει κανένα που τα διαβάζει. Το 1% και πολύ λέω. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να το έχουμε μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Αν κάποιος θέλει χαρτί να το ζητάει. Α, αλλά εγώ πραγματικά όποτε παίρνω ε, το αντίγραφο σε χαρτί το πετάω στο είναι και κατευθείαν. Είναι και αυτό ένα, μια περιττή δαπάνη. Και άλλα πράγματα μπορώ να πω για το χαρτί. Ε, για το ή ε, μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα χρησιμοποιώντας λιγότερο χαρτί. Ε, έχουμε την ε, διάταξη ολομέλειας για τέσσερις μέρες, έχουμε την προσωρινή ημερησία διάταξη, έχω την πλήρη μερίσια διάταξη, έχουμε την ε, συνοπτική ημερησία διάταξη, πολλά έγγραφα, τα οποία πραγματικά χρειάζεται κάποιος να, τα παράγει ε, και, και αυτό είναι σπατάλη ανθρώπινου δυναμικού. Ας το σκεφτείτε. Επίσης μπορούμε να συνεχίσουμε το πάγωμα ε, των επιδομάτων των ε, βουλευτών. Αυτό βέβαια θα το αποφασίσουμε εμείς, τα μέλη, πρόκειται για μια πολιτική απόφαση. Ε, ο πληθωρισμός ίσως θα μπορούσε επίσης να σας βοηθήσει. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός τον επόμενο χρόνο θα είναι 1,1%. Αυτό επίσης θα βοηθήσει στη ε, ε, διατήρηση του κόστου σε χαμηλά επίπεδα. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για όλα όσα έχετε κάνει τα τελευταία πέντε χρόνια και ελπίζω ότι μαζί θα καταφέρουμε ακόμα περισσότερα τα επόμενα χρόνια. Και κάτι ακόμα. Χτες έλαβα μια παρουσίαση από την βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου. Το 2007 είχαμε προτείνει διαχείριση γνώσης από το Κοινοβούλιο και αυτό το πετύχατε, το καταφέρατε. Τώρα τα ε, μέλη μπορούν να, να αναζητούν πληροφορίες πολύ γρήγορα. Θέτεις ένα ερώτημα και μέσα σε τρεις ώρες παίρνει την απάντηση. Αυτό είναι εξαιρετικό. Είναι μια πραγματική ευκαιρία για τους συναδέλφους και πρέπει να υποφεληθούν από αυτή τη δυνατότητα. Ε, μπορεί κανείς να λαμβάνει ειδοποιήσεις όταν εμφανίζεται καινούρια πληροφορία που ενδιαφέρει. Μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα. Πραγματικά θέλω να συγχαρώ το Γενικό Γραμματέα για όλα όσα έχει κάνει αυτά τα χρόνια. Ελπίζουμε θα συνεχίσουμε. Merci. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Δεπρά έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και το Γενικό Γραμματέα. Σας ζητώ συγγνώμη, διότι σε λίγα λεπτά θα πρέπει να αποχωρήσω. Έχω μια άλλη υποχρέωση στις 12.30, δεν μπορώ να καθυστερήσω. Απευθυνόμενος λοιπόν στο Γενικό Γραμματέα να του πω ότι τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσίασή του, πολύ καλά δοδημένη, πάρα πολύ σαφής. Όσον αφορά τις προτεραιότητες κύριε Πρόεδρε, ήδη είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε τις προτεραιότητες Νομίζω ότι πάρα πολύ πάντως συμφωνούμε για τις πιο σημαντικές προτεραιότητες οι οποίες εσείς θίξατε κύριε Γενική Γραμματέα. Η ασφάλεια, όλοι συμφωνούμε επ' αυτού. Η ασφάλεια των κτηρίων, η πρόσβαση στα κτίρια. Καθώς επίσης και η εξωτερική ασφάλεια που εξαρτάται με τις διαπραγματεύσεις που έχουμε με τα κράτη-μέλη. Επομένως, σας ενθαρρύνουμε να ακολουθήσετε όντως αυτό το δρόμο. Αναφερθήκατε όμως επίσης και στην πληροφορική. Όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν βρίσκεται στο υψηλότερο δυνατό επαγγελματικό επίπεδο. Νομίζω δηλαδή ότι στον τομέα αυτό θα πρέπει να γίνουν αναλύσεις, μελέτες και κάποιε αναγκαίε τροποποιήσει για να βελτιωθεί η κατάσταση. Συμφωνώ πάντως μαζί σα, κύριε Γενική Γραμματέα, ότι πρέπει να αυξήσουμε τι ικανότητέ μα όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Νομίζω υπήρχε μια κάποια συνένεση ήδη στα μέλη εδώ πέρα της Επιτροπής μας όταν παρουσίασα για πρώτη φορά το προσχέδιο εγγράφου εργασίας, όταν είπα συγκεκριμένα ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την δυνατότητα των Ευρωπαϊκών Επιτροπών να ασκούν πραγματικά έλεγχο. Και ως προς αυτό κάνατε μια πολύ σωστή πρόταση κύριε Γενική Γραμματέα. Θεωρώ ότι πρόκειται μια, για μια πάρα πολύ σημαντική προτεραιότητα. Να καταφέρουμε να ενισχύσουμε την διοικητική υποστήριξη προς ευρωβουλευτές προκειμένου αυτοί να ασκούν τον, το ελεκτικό τους έργο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χαιρετίζω επίσης τα όσα είπατε σχετικά με τις καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους ευρωβουλευτές. Όντως, είμαστε ορισμένοι ευρωβουλευτές καταδικασμένοι να εργαζόμαστε σε κάποια πολύ μικρά γραφεία με τον βοηθό μας δίπλα. Ξέρετε ότι δεν είναι δυνατόν να εργαστούμε σε αυτές τις συνθήκες, δεν μπορούμε να δεχθούμε επισκέπτες, δεν μπορούμε να διοργανώσουμε μια συζήτηση εργασίας, μια συνάντηση εργασίας στα πλαίσια των πολύ μικρών αυτών γραφείων. Θα ήθελα λοιπόν να βοηθήσουμε τους 300 αυτούς κακόμερους ευρωβουλευτές, οι οποίοι παραμένουν ακόμη σε κάποια πολύ μικρά γραφεία. Επίσης, η πρότασή σας να έχουμε κάποιες ε, συγκεκριμένες νέες μορφές για τον εξοπλισμό, ε, κάποια συγκεκριμένα πρότυπα για την επίπλωση και αυτό είναι πολύ ε, σημαντικό. Τώρα η αύξηση, 2,93%. Η αύξηση αυτή στην οποία αναφερθήκατε Ξέρετε ότι η συνολική αύξηση του προπολογισμού του Κοινοβουλίου τελικά θα εξαρτηθεί από τις επιπλέον ανάγκες, από, την, από τον τιμάριθμο, καθώς επίσης και από την εξοικονόμηση που θα αποφασίσουμε να κάνουμε. Όπως το είπατε και εσείς κύριε Γενική Γραμματέα, ακόμα σε πολλούς τομείς μπορούν να γίνουν σημαντικές εξοικονομήσεις. Συνεπώς, δεν θα τοποθετηθώ σήμερα για το αν θα πρέπει να μείνουμε στο 2,9% ή στο 3%. Δεν απόκειται άλλωστε σε μένα να το πω, δεν χρειάζεται να πάμε πάντως τόσο μακριά. Ωστόσο υπάρχει ένα λεπτό, ένα ευαίσθητο θέμα το οποίο θα ήθελα να θίξω αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά την αύξηση των αποζημιώσεων για τη γραμματεία. Θα υποβάλω μια πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να γίνουν κάποιοι έλεγχοι, μάλλον έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι, κάποιες έρευνες για τις αποζημιώσεις αυτές και καταλήγουμε τελικά στο συμπέρασμα ότι ε, ορισμένοι συνέδελφοι και συγκεκριμένα σε κάποιες πολιτικές ομάδες ε, χρησιμοποιούνται πάρα πολύ τοπική βοηθή, ζητούν ιδιαίτερα σημαντική τοπική υποστήριξη και όχι τόσους πολλούς πιστοποιημένους ε, ε, βοηθούς. Και αυτό γιατί πολλές φορές δεν έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχουν την απαραίτητη αυτή υποστήριξη που τους επέτρεπε να λειτουργούν πλήρως ως ευρωβουλευτές. Επομένως, το επίδομο γραμματείας το οποίο προτείνεται να αυξηθεί θα αποτελέσει θα το ζητήσω τουλάχιστον αυτό αντικείμενο συζήτηση τη δική μα επιτροπή, προκειμένου να έχουμε πιο αυστηρού κανόνε ω προ αυτό. Θα μπορούσαμε δηλαδή να κινηθούμε προς μία αύξηση. Για τους πιστοποιημένους, για παράδειγμα βοηθούς, θα μπορούσε να υπάρχει μία, μία αύξηση για τους διαπιστευμένους με συγχωρείτε βοηθούς. Αλλά νομίζω ότι σε κάποιες άλλες περιπτώσεις θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες εξοικονομήσεις. Και αν προβλέπουμε συνεχώς αυξήσεις τελικά πού θα θέσουμε το όριο. Μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Νομίζω ότι γενικότερα η κατάσταση είναι κάπως δυσανάλογη και νομίζω ότι δεν μπορούμε να μείνουμε σε τέτοιους αριθμούς. Καταλαβαίνετε ότι ε, η ίδια εξοπιστία μας απέντη στην κοινή γνώμη τίθεται ένα αφιβόλο αυτή τη στιγμή. Κάθε φορά που μιλάμε για τη διάκριση αυτή που γίνεται ανάμεσα σε τοπικούς βοηθούς και διαπιστευμένους βοηθούς. Θα ήθελα λοιπόν να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για αυτό το ζήτημα, γιατί το να αυξήσουμε απλώς το επίδημα το οποίο προβλέπεται για την γραμματεία, νομίζω ότι ουσιαστικά για τη γραμματιακή υποστήριξη δεν μας οδηγεί στο σωστό δρόμο. Πρέπει να θέσουμε κάποιους κανόνες και να γίνει μια συζήτηση προς αυτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, πρέπει να αποχωρήσω. Παρακαλώ θα σας έδινα τους άλλους τον λόγο και θα πρέπει να επιταχύνουμε τώρα λίγο και τη συζήτηση. Μπορείτε να περιοριστείτε οι υπόλοιποι ομιλητέ σε δύο λεπτά αναπαρέμβαση. Ο κύριος Τάραντ έχει το λόγο. ευχαριστώ να περιοριστώ στα δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Βέλε για την ε, παρουσίαση αυτή όσον αφορά τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να κάνω κάποιες προτάσεις και μια πρόταση με τη μορφή ερώτησης. Με ποιον θα μπορούσα εγώ να συνεργαστώ στα πλαίσια της γραμματείας προκειμένου να καταφέρω να χρησιμοποιώ λογισμικό open source. Γιατί διαφορετικά ουσιαστικά πληρώνουμε τον Bill Gates ο οποίο είναι πολύ καλό κύριο ενδεχομένω και έχει και πολύ σημαντικό έργο φιλανθρωπία, αλλά θα μπορούσαμε να το κάνουμε και εμεί αυτό. Μπορώ λοιπόν εγώ ω Ευρωβουλευτή να έρθω σε επαφή με κάποιον προκειμένου να μπορώ να χρησιμοποιώ αυτό το λογισμικό, το ανοιχτό λογισμικό. Δώστε μου γι' αυτό μια απάντηση κύριε Γενική Γραμματέα. Δεύτερον, επί της διαδικασίας θα μπορούσατε ακριβώ να μου πείτε το Προεδρείο είναι αυτό το οποίο θα αποφασίσει για την κατάσταση των προβλέψεων, για τα συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα. Έτσι δεν είναι. Θα μπορούσε όμως στη συνέχεια η δική μας Επιτροπή να τροποποιήσει αυτή την κατάσταση προβλέψεων ή ο τελικός λόγος τελικά νίκη στο Προεδρείο. Όσον αφορά επίσης τις γλώσσες, το αναφέρατε κι εσείς αυτό. φτυχώς δεν έχουμε σήμερα Εστονούς διερμηνείς, άρα μπορώ ανοιχτά να μιλήσω σήμερα, διαφορετικά θα με λιθοβολούσανε. Κατά την άποψή μου, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μία τροποποίηση της ε, συνθήκης του κανονισμού έτσι ώστε να έχουμε γαλλικά, γερμανικά, πολωνικά ως βασικές γλώσσες, τα ισπανικά επίσης ως μελλοντική γλώσσα των ΗΠΑ και πέρα από τις υποχρεωτικές αυτές γλώσσες, αν κάποιοι σε μια εκλογική περιφέρεια είναι αρκετά νόητοι ώστε να, μην, να εκλέξουν κάποιον που δεν μπορεί να μιλήσει καμία από τις πέντε αυτές γλώσσες, τότε θα μπορούσαμε ενδεχομένω να προσλάβουμε έναν βοηθό, ο οποίος θα μπορούσε να μπει στην καμπίνα και να μεταφράσει. Κατά αυτόν τον τρόπο θα εξοικονομούσαμε πάρα πολλά χρήματα. Πέρασαν και τα δύο μου λεπτά. Σας ευχαριστώ. Madame Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς, ε, συμφωνώ όλα όσα λέγονται για τη βελτίωση στις εισόδους. Η κατάσταση είναι τόσο λυπηρή. Αυτές οι περιστραφόμενες πόρτες που έχουμε ούτε τεχνικά είναι καλές. Σήμερα το πρωί είδα στις 9 παρατέταρτο όταν ήθελε τόσος κόσμος μέσα γίνονται ουρές αυτές οι περιστραφόμενες ε, πόρτες. Δεν μπορεί να περάσει κανείς. Όταν τις φτιάξαμε αυτές τι πόρτες δεν υπολογίζαμε πόσο κόσμος θα έπρεπε να τι χρησιμοποιεί και για λόγους ασφαλείας αλλά και για, και για λειτουργικούς λόγους. Πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση. Οπότε ερώτηση. Δεν μπορούμε να δούμε τι κάνουν τα άλλα κοινοβούλια, πώς επιλύονται αυτά τα προβλήματα. Γιατί έχουμε πολύ σύγχρονα συστήματα. Άλλα κοινοβούλια βέβαια μπορεί να έχουν πεπαλαιωμένα, αλλά σίγουρα κάποια κοινοβούλια έχουν ε, σύγχρονα συστήματα από τη μία να δείχνουν ότι θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί και διαφανείς αλλά ότι θέλουμε να διασφαλίσουμε και την ε, ασφαλεία μας ούτως ώστε όποιοι δεν δικαιούνται να μην μπορούν να εισέλθουν και να είμαστε ασφαλείς ε, από ενδεχόμενο επίθεσης. Γιατί μια επίθεση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο έξω από το κτίριο και το εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να προσφέρει ένα κάποιο επίπεδο ασφάλειας, αλλά να είναι ελκυστικό. Για τα κτίρια, επίσης, μια παράκληση. Εφόσον θα ανακαινήσουμε το Polaris Risk Park, αυτή τη στιγμή έχουμε πλέον και σύγχρονα συστήματα διαχείρισης του ποσίμου ύδατος. Αυτή τη ε, στιγμή ε, δαπανούμε εκατομμύρια και χρησιμοποιούμε πολλές χιλιάδες μπουκάλια διότι το νερό της βρύσης δεν είναι παρκώς καλό. Έχουμε σύγχρονα συστήματα διαχείρισης του ύδατος. Θα μπορούσαμε λοιπόν να τα εγκαταστήσουμε ούτως ώστε το νερό που περνάει από τη μία να μην καταστρέφει τους σωλήνες και από την άλλη να είναι τόσο καλής ποιότητας που να μπορούν όλοι να το πιούν. Και τελευταίο, τα εστιατόρια. Είπατε ότι πρέπει να έχουμε πάνω από μία επιχείρηση, δηλαδή όχι μόνο τη οντέξω. Πολύ θετικό. Το κτίριο ε, ε, Park δεν έχει καν τη δυνατότητα να ζεστάνει κανείς κάτι ή να το βάλει σε ένα ψυγείο για να μπορεί να το φάει αργότερα. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν κάποιες τέτοιες εγκαταστάσεις ε, για ένα κτίριο που χρησιμοποιούν τόσες χιλιάδες άτομα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριο Βάλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος, ε, γιατί όμω δεν έχουμε πολύ χρόνο. Μία παρατήρηση όσον αφορά την αύξηση του προπολογισμού κατά 3%. Νομίζω την υπερβολική αύξηση αυτή, ιδίω σε μια περίοδο στασιμότητα ύφεση και ξέρετε ότι πολλά κράτη-μέλη χρειάστηκε να κάνουν σημαντικέ περικοπέ σε μισθού, συντάξει και άλλε κοινωνικέ παροχέ και δημόσιε δαπάνε. Μου φαίνεται λοιπόν παράλογο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην το λαμβάνει αυτό υπόψη και να προβλέπει αύξηση του προπολογισμού. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δύσκολα θα γίνει αποδεκτό από άλλα κράτη-μέλη. Δεύτερον, πέρασαν οι ευρωπαϊκές εκλογές, είναι πλέον μακριά. Οι δαπάνε, οι σχετικέ όσον αφορά την προκλογική εκστρατεία, ποιε ακριβώ ήταν, δεν μπορούσα να καταλάβω το σημείο αυτό. Ενδεχομένω θα μπορούσατε να μου δώσετε περαιτέρω διευκρινήσει. Επίση, λέγεται ότι ορισμένε πολιτικέ ομάδε θέλουν να αιτηθούν αύξηση του επιδόματο γραμματιακή υποστήριξη ε, και ξέρω ότι εμείς ε, επιτελούμε ένα πολύ σημαντικό έργο, έχουμε πολύ σημαντικές ευθύνες, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δοθούν ε, πάλι να δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το σωστό παράδειγμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιες αυξήσεις. Τώρα, για την αποζημίωση αυτή στην οποία αναφερθήκατε της γραμματικής υποστήριξης ενδεχομένως θα μπορούσατε να μας δώσετε εδώ πέρα κάποιες περισσότερες πληροφορίες και να υπάρχει και περισσότερη διαφάνεια και για τις ταξιδιωτικέ δαπάνες θα μπορούσαμε να είχαμε μια κάποια σύμβαση, συμφωνία με τι αεροπορικέ εταιρείε, γιατί αυτό που βλέπουμε πολύ συχνά είναι ότι είναι πολύ ψηλέ αυτέ οι δαπάνε. Κάθε φορά που οι δικοί μου συνεργάτε, για παράδειγμα, μου κλείνουν διάφορα εισιτήρια, βλέπω ότι η τιμή των εισιτηρίων είναι πάρα πολύ ψηλή. Ενδεχομένω λοιπόν ήταν σκόπιμο να δούμε αν μπορούμε να περιορίσουμε αυτέ τι δεξιωτικέ δαπάνε. Εγώ πολύ συχνά ταξιδεύω βέβαια στην οικονομική θέση και ελπίζω ότι αυτό κάνουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, ότι δεν ταξιδεύουν αναγκαστικά στην διακεκριμένη θέση. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της ασφάλειας, από όσο ξέρω, στο Στρασβούργο καλυπτόμαθα από τις ε, γαλλικές αρχές. Στο Βέλγιο όμως, καθότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα φέρουν ένα μεγάλο μέρος της δαπάνης, νομίζω ότι θα πρέπει ε, να δούμε τελικά πώς μπορούμε τα χρήματα αυτά τα οποία εμείς ε, χρησιμοποιούμε και επενδύουμε να χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και συνεργασία με τις βελικές αρχές. Επίσης, η θέρμανση, ο εξαιρισμός ε, πολύ συχνά δεν λειτουργούν πολύ σωστά και εκεί πέρα μπορεί να γίνουν κάποιες βελτιώσεις όσον αφορά το νερό, ας χρησιμοποιούμε λιγότερα πλαστικά μπουκάλια, 30 εκατομμύρια ευρώ συνολικός υπροπολογισμός για το σπίτι της ευρωπαϊκής ιστορίας. Πώς θα διαχειριστούμε τις δαπάνες αυτές, ποια θα είναι η κατανομή ανά έτος. Δεν ξέρω αν οι Ευρωπαίοι πολίτες θα ενέκριναν ποτέ τέτοιε δαπάνες. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε κύριε Βάλη. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Γενικό Γραμματέα για όσα είπε για την ε, ευελιξία που είναι αναγκαία για τον προπολογισμό. Υπάρχουν ε, συνάδελφοι οι οποίοι εργάζονται εντατικά και που παίρνουν σοβαρά τη δουλειά τους και υπάρχει και το αντίθετο. Και γι' αυτό είναι πολύ διαφορετικές οι ανάγκες των συναδέλφων. Άλλοι εργάζονται πολύ, άλλοι πολύ λίγο. Και υπάρχει όντως ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων που όντως δουλεύουν πολύ. Γι' αυτό ο κάθε βουλευτής πρέπει ο ίδιος να αποφασίζει πώς θα χρησιμοποιήσει το επίδομα γραμματείας και ποιους θα προσλάβει. Όποιος ε, εργάζεται λιγότερο και δεν χρειάζεται συνεργάτες μπορεί να βοηθήσει το κοινοβούλιο να κάνει εξοικονομήσεις και όποιος ε, προσλαμβάνει ανθρώπους χαμηλού επίπεδου και τους ε, πληρώνει λίγα και αυτός μπορεί να βοηθήσει σε εξοικονομήσει το κοινοβούλιο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ευέλικτοι. Φυσικά να υπάρχει ένα νοτοτόριο μέχρι ποιο ποσό μπορεί να πληρώσει κανείς για βοηθούς, ακόμη και αν είναι υψηλωτά του επίπεδου. Και είναι σαφές ότι αν κάποιος θέλει να προσλάβει έναν πρώην Υπουργό Οικονομικών ή Εξωτερικών, θα ήταν καλό να υπάρχει με κάποια ευελιξία. Αυτό είναι το αποφασιστικό. Έχουμε όλοι τα διάφορα ηλεκτρονικά μέσα, άρα όλοι τα χρησιμοποιούμε και μας βοηθούν να έχουμε πολύ καλή ποιότητα εργασίας. <clears throat> Θα μπορούσε αυτό να είναι χρήσιμο και για την είσοδο στο κοινοβούλιο. Το προσωπικό στο Αυστραλιανό Κοινοβούλιο, για παράδειγμα, <clears throat> έχει δυνατότητα μέσω των smartphones να δει αν κάποιος είναι ευρωβουλευτής και επίσης να δει και τι άλλες κατηγορίες ε, ατόμων, λομπίστες ή άλλοι θέλουν να μπουν στο κτίριο. Πρέπει επίσης να πλουστεύσουμε τα ταξιδιωτικά μας έξοδα. Άκουσα ότι ορισμένες φορές οι έλεγχοι των ταξιδιωτικών εξόδων κρατάνε περίπου ένα χρόνο μέχρι να γίνει επιστροφή των εξόδων. Δεν είναι δυνατόν να κρατάνε τόσο πολύ. Πρέπει να είναι πιο ταχύς ο έλεγχος και η επιστροφή. Επίσης για τα ταξίδια. Οι ευρωβουλευτές πρέπει να έχουν επίσης κάθε δικαίωμα όταν κάνουν ταξίδια στον κόσμο να έχουν τουλάχιστον ένα συνεργάτη μαζί τους να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Ευχαριστώ πολύ, λέω ο Η κυρία Γκαρθιαδάβαλ. Δύο ερωτήσεις μόνο γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας σχεδόν. Είπε ο Γενικός Γραμματέας γιατί μίλησε για την ενίσχυση ε, ή τη δημιουργία υπηρεσιών για τις κατεξιοδότηση πράξεις που θα μας φτάσουν και μίλησε και για την αύξηση, βελτίωση της τεκμηρίωσης και υποστήριξης προς τους ε, βουλευτές. Ε, για πόσο προσωπικό μιλούμε. Γιατί ε, έτσι κι αλλιώς πρέπει να κάνουμε μείωση του προσωπικού στις υπό, στα υπόλοιπα όργανα για Δεύτερον, το θέμα του παιδικού σταθμού του Κοινοβουλίου. Ξέρουμε ότι υπάρχουν τεράστιες ε, ε λίστες αναμονής. Ε, ε, θα θέλατε να μου πείτε τι, τι εξέλιξη έχουμε σε αυτό το μέτωπο. Merci. Monsieur Gaillard, derrière intervenant. Ο κύριος Γκάλερ, τελευταίος. Πολύ σύντομα. Γκάιερ, συγγνώμη. 3% νομίζω ότι το ποσό αυτό του 3% δεν είναι και λίγο, αλλά δεν είναι κατά ανάγκη και επαρκές. Θα ήθελα να μας πείτε τι ποσοστό αυξήσεων ε, προβλέπετε για παράδειγμα για το ηλεκτρικό στο Βέλγιο. Το δεύτερο είναι κάτι που το είπε και ο Πάουλ Ρούμπιχ μόλις τώρα. Αν όντως ισχύει ότι κάποιοι βουλευτές έχουν μηδέν βοηθούς της Βρυξέλλες και 40 στην εκλογική τους περιφέρεια, νομίζω ότι είναι παράνομη χρηματοδότηση του κόμματος αυτό. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να τα κάνει όλα μόνο του εδώ στις Βρυξέλλες και να έχει 40 άτομα στην χώρα του. Πρέπει να τα εξηγήσει κανείς αυτά στους ε, εκλογείς πώς τα κάνει αυτά. Νομίζω ότι θα ήταν ε, σκόπιμο να υποχρεούνται οι βουλευτές να έχουν συνεργάτες στις Βρυξέλλες και αν δεν έχουν να τους μειώνεται το επίδομα γραμματείας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γενική Γραμματέα, αυτές ήταν οι ερωτήσεις και παρατηρήσεις. <clears throat> σας παρακαλώ να είστε σύντομος στις απαντήσεις σας. Θα επανέλθουμε φυσικά επί ορισμένων θεμάτων. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Αλλά επειδή υπήρξαν πολλές ερωτήσεις, ε, δεν ξέρω πόσο σύντομο θα είναι. Στις ερωτήσεις του κυρίου Μάνκα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα του ελέγχου που κάναμε για τα κτίρια, την υπηρεσία κτίριων. Υπόθηκε ότι πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα για τη συντήρηση των κτίριων. Αυτό έγινε. Γιατί αν δεν κάναμε αυτή την προσπάθεια να ελέγξουμε πού πρέπει να κάνουμε συντήρηση, δεν θα είχαμε ανακαλύψει ότι είναι σαθροί η οροφή και θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες αυτό. Νομίζω ότι σε αυτή την περασμένη πενταετία <clears throat> καταφέραμε να περάσουμε από την αντίληψη του ότι έχουμε καινούργια κτίρια που δεν χρειάζονται πολύ συντήρηση, στην αντίληψη ότι πρέπει να ασχολούμεθα και με τα νέα κτίρια και με την μίσθωση νέων κτίριων και με τις επισκευές και για το κόστος. Μπορώ να σας πω ότι ε, εκτελέσαμε πολύ μεγάλα προγράμματα οικοδόμησης κτηρίων και όλα αυτά χωρίς υπέρβαση. Αυτό και για το τεράστιο κτίριο Κόντραντ Αντενάρ στο Λουξεμβούργο. Δεν έχει τελειώσει ακόμη, πρέπει να είμαι λοιπόν ε, προσεκτικός. Αλλά επειδή έχουμε και καλή βοήθεια από συμβούλους, πιστεύω ότι και εδώ δεν θα υπάρξει υπέρβαση. Τα τελευταία χρόνια είπαμε ότι η στρατηγική μας είναι θέλουμε να κάνουμε και καινούργια πράγματα. Δεν θέλουμε να μείνουμε στην παρούσα κατάσταση, αλλά ότι ορισμένα πρέπει να γίνουν και με εξοικονομήσεις. Δηλαδή να εξοικονομήσουμε από παλιές δαπάνες για να μπορέσουμε να έχουμε νέες δαπάνες. Είχαμε ορισμένες λοιπόν θετικές και ορισμένες αρνητικές προτεραιότητες. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε περιθώρια ελιγμών που αλλιώς δεν θα τα είχαμε αν δεν είχαμε αυτή την ευέλικτη στρατηγική. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Επιτροπή Προπολογισμών γιατί πάντα μας βοήθησε όταν αγοράσαμε για παράδειγμα κτίρια πάντα μας έδωσε τη δυνατότητα οποιαδήποτε πλεονάσματα να τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε δαπάνες ε, νωρίτερα από ό,τι προεβλέπετο για να γλιτώσουμε τόκους. Για παράδειγμα, εάν δώσουμε 50 εκατομμύρια νωρίτερα, μπορούμε να γλιτώσουμε 16-17 εκατομμύρια σε τόκους κατά την διάρκεια ε, αποπληρωμής των κτηρίων. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να τηρήσουμε αυτή την στρατηγική που ήταν δυνατή επειδή είχαμε μέσο και μακροπρόθεσμη στρατηγική. Έχετε δίκιο ότι χρησιμοποιούν πολύ διαφορετικά οι βουλευτές τη δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων και αυτό δημιουργεί κόστος και στην Κομισιόν και μας δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένα στοιχεία. Αναφερθήκατε στην ε, μετάφραση των τροπολογιών. Στην προηγούμενη διαδικασία έγκρισης προπολογισμού που είπαμε ότι σε επίπεδο επιτροπής θα μεταφράζονται μόνο στις γλώσσες των μελών της Επιτροπής. Γιατί πολλές τροπολογίες δεν πάνε τελικά στην Ολομέλεια. Έτσι ήδη έχουμε κάποιες ε, οικονομίες. Μόνο στις γλώσσες που χρειάζεται μεταφράζονται σε επίπεδο επιτροπής οι τροπολογίες. Αυτή η σκέψη να γίνεται μόνο ανάλογα με το τι αιτήματα έχουν υποβληθεί, αυτό μας οδήγησε στο να δούμε επίσης ότι και τα αναλυτικά, αναλυτικά πρακτικά τη Ολομέλεια δεν μεταφράζονται πλέον συστηματικά και κανεί βουλευτή δεν μοιάζει να διαμαρτύρεται ότι δεν έχει πια αυτή τη δυνατότητα και αυτό οδήγησε σε οικονομίε 10 εκατομμυρίων. Επίση, τα πρακτικά των ε, επιτροπών δεν τυπώνονται, υπάρχουν μόνο ηλεκτρονικά. Αυτό πρέπει να ισχύει γενικά στο Κοινοβούλιο Ήδη ε, τα τελευταία πέντε χρόνια μειώσαμε στο 50% την κατανάλωση χαρτιού. Θα μπορούσαμε όμως ε, να έχουμε ένα επιπλέον 10% μείωση της κατανάλωσης ε, χάρτου. Ο κύριος Ντεπρέ είπε ότι συμφωνεί με, την, με τις ενέργειές μας για την ασφάλεια και ότι πρέπει να βελτιώσουμε την κυβερνοασφάλεια. Αλλά δεν είναι πολύ απλό όταν θέλουμε να έχουμε παντού συνδεσιμότητα με τα πιο διαφορετικά μηχανήματα και τις πιο διαφορετικές ε, προδιαγραφές. Πρέπει φυσικά να γίνουν επενδύσεις για να το επιτύχουμε και αυτό. Ευχαριστώ πολύ για την στήριξή σας. <clears throat> Ότι οι επιτροπές πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στην επίβλεψη όλων αυτών και για τις καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους βουλευτές όπως σας είπα Περιμένουν ακόμη 300 βουλευτές άλλο ένα γραφείο, επίσης και πιο ευέλικτη και σύγχρονη <clears throat> διαμόρφωση και διαρρύθμιση των γραφείων. Αναφέρθηκαν οι κανόνες για τους ε, βοηθούς στις εκλογικές περιφέρειες. Πρέπει να ελέξουμε τα στοιχεία πιο συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ ευέλικτοι Ίσως να είμαστε υπερβολικά ευέλικτοι στο τι επιτρέπουμε. Ίσως θα ήταν καλό να δούμε τις λεπτομέρειες. Ο κύριος Ταρά αναφέρθηκε στο λογισμικό ανοιχτή πηγής, open source. <clears throat> ναι, έχουμε μια σειρά από τέτοια λογισμικά που αξιοποιούμε. Ο Γενικός Διευθυντής ε, Πληροφορικής, ο κύριος Βιλέλα, ασχολείται με τα θέματα αυτά συμμετέχει σε συζητήσεις για τα θέματα αυτά είναι στη διάθεσή σας. Για τη διαδικασία του προπολογισμού. Το Προεδρείο αποφασίζει τις καθεντήρες γραμμές μετά το προσχέδιο, όπως υποθέτω θα γίνει σε 9 Μαρτίου, και μετά επανερχόμεθα στην Επιτροπή Προπολογισμών, όπως κάθε χρόνο, και προσπαθούμε και καταλήγουμε σε μια συμφωνία που εγκρίνεται από το Προεδρείο και την Επιτροπή Προπολογισμών. Θέλουμε λοιπόν να καταλήξουμε σε ένα κείμενο που να βρίσκει και τις δύο αυτές αρχές σύμφωνες και που να μας επιτρέπει να χρηματοδοτήσουμε τις, ε, τη λειτουργία μας. Τώρα για τις γλώσσες δεν θα πω τίποτα, εργαζόμαστε με βάση τις συνθήκες, όπως ισχύουν. Όσο έχουμε αυτές τις συνθήκες θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να είναι όσο δυνατόν πιο αποτελεσματικές οι υπηρεσίες μας για να εγγυώνται την πολυγλωσσία. Η κυρία Χολμάιρ αναφέρθηκε στις ε, περιστρεφόμενες πόρτες. Θα τι αλλάξουμε του επόμενους μήνε Είναι παλιέ. Σίγουρα δεν είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Για τις πόρτες δεν θα περιμένουν μέχρι του χρόνου. Οι πόρτες τους επόμενους μήνε θα αλλάξουν. Έχουν γίνει ήδη προκήρυξεις. Η νέα διαμόρφωση των εγκαταστάσεων ασφάλειας Θέλουμε να είναι στο επίπεδο τεχνολογίας που υπάρχουν των ε, καταστάσεων της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Είναι τελευταία που διαμόρφωσε τα κτίρια της, με τις αναγκαίες φυσικά προδιαγραφές ασφάλειας. Αυτό θα είναι το πρότυπό μας. Άρα θα σημειώσουμε πιστεύω ουσιώδη πρόοδο. Και θα πρέπει να θέσουμε και το ερώτημα ποιος θα περνάει από ποια πόρτα όλοι από όλες τις πόρτες ή ειδικέ πόρτες για κάθε κατηγορία εισερχομένων. Αυτό όμως είναι πάντα λεπτό θέμα. Για την συντήρηση του Polaris Pack, σύγχρονη διαχείριση ύδατος, σύγχρονα μαγειρία, βεβαίως. Πρέπει να δούμε εάν θα μείνει ως έχει, ως διαμόρφωση το Polaris Pack ή αν του λείπουν κάποιες λειτουργίες, μήπως η συντήρηση θα είναι μια ευκαιρία για να βελτιώσουμε τις λειτουργίες. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις αίθουσες συνεδριάσεων, αν μπορούμε να διαμορφώσουμε κάποιες αίθουσες για τριμερείς διαλόγους, όπου δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κατάλληλες αίθουσες. Ο κύριος Βάλλη αναφέρθηκε στο 3%. Στον τομέα του προσωπικού μελετήσαμε τι επιπτώσεις έχει το σύστημα προαγωγών μας, βαθμοί και κλιμάκια και είδαμε και τι συμβόλαια έχουμε που πολύ συχνά προβλέπουν ε, τιμαριθμικές αναπροσαρμογές. Υπάρχουν δηλαδή θέματα που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Για το 16 δεν έχουμε εκλογικέ δαπάνες. Αυτό προσπάθησα να πω. Δεν έχουμε για το 16. Εδώ λοιπόν μπορούμε να προωθήσουμε άλλες χρηματοδοτήσεις για το επίδομα γραμματείας είπα είναι πολιτικό το θέμα. Αλλά είναι σημαντικό να λαμβάνουν συμβουλές και στήριξη οι βουλευτές από διάφορες πηγές διότι δεν είναι δυνατόν να εξαρτώμεθα από λόμπι για υψηλής εξειδίκευσης νομοθετικά θέματα διότι βεβαίως έχουν πολλές συμβουλές να μας δώσουν τα λόμπι αλλά δεν είναι κατά ανάγκη να μερόληπτες. Πρέπει λοιπόν το Κοινοβούλιο και οι βουλευτές να μπορούν να λαμβάνουν ε, ενημέρωση και στήριξη από διάφορες πηγές. Βεβαίως το βαλικό κράτος αναγνωρίζει την ευθύνη του για μας. Έτσι το διαπιστώσαμε από τα μηνύματα που λάβαμε τους τελευταίους μήνες. Το σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας τώρα. Έχουμε μια συμφωνία με την Επιτροπή Προϋπολογισμών από το 2012 για τις επενδύσεις, μπορεί να γίνει το κόστος της επένδυσης, τα τρέχοντα έξοδα. Σε σημερινές τιμές είχαν καθοριστεί σε 12,5 εκατομμύρια τα λειτουργικά τρέχοντα έξοδα. Πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι έχουμε διαπιστώσει τόσο μεγάλη προσέλευση στο παρλαμεντάριο που έχουμε φτάσει στα όρια. Είχαμε πάνω από ένα εκατομμύριο επισκέπτες στο παρλαμεντάριο. Είναι τόσο μεγάλη προσέλευση ιδιαίτερα από πλευρά ε, σχολείων που θέλουν να παίξουν αυτό το παιχνίδι ρόλων, ορισμένε περιόδου αρχέ του χρόνου χρειάστηκε να αρνηθούμε τρει από τι τέσσερι ε, αιτήσει επισκέψεων που λάβαμε. Αυτό λοιπόν ε, σημαίνει πω καλή είναι και η πρωτοβουλία. Κύριε αναφέρατε τα ανώτατα ποσά για τις αποδοχές. Υπάρχουν συστάσεις του Προεδρείου που έχουν νομίζω εφαρμοστεί έχουν συζητηθεί για τη σύγχρονη τεχνολογία στον τομέα της ασφάλειας και σημείωσα και αυτό που ότι πρέπει να μπορούν να ταξιδέψουν και οι βοηθοί. Η κυρία Κουάρδια Θάβαλ μίλησε για τις ε, κατεξολόγηση κατ εξουσιοδότηση πράξης. Θα τηρήσουμε τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει μείωση του προσωπικού 1% το χρόνο του οργανογράμματος. Με βάση το οργανόγραμμα της 1ης πρώτου 12. Αυτό θα το κάνουμε. Θα μειώσουμε τις θέσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αρχές, η αρχή του προπολογισμού, αν υπάρχει επίγουσα ανάγκη, δεν θα πρέπει να έχει δυνατότητα για κάποιες υπηρεσίες να προβλέψει επιπλέον θέσεις. Το κάναμε και στους προηγούμενους προπολογισμούς, για παράδειγμα για την πληροφορική, όπου επίση επαναφέραμε εντό του οργανογράμματο κάποιε υπηρεσίε, υπάρχει δυνατότητα, πρέπει να αξιοποιείται προσεκτικά, σύνετα, αλλά για τις κατεξοδότηση, πράξη και την ασφάλεια θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Τέθηκε ένα ερώτημα για το δεύτερο νηπιαγωγείο. Έχουμε περίπου 50 άτομα σε λίστα αναμονής. Θέλουμε να έχει τέσσερις τάξεις το νηπιαγωγείο για να ικανοποιήσουμε αυτά τα αιτήματα. Ο κύριος Γκάια ρώτησε ποια είναι η βάση της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής έχει να κάνει με τις αυξήσεις ε, των μισθών λόγω των προογών και την ε, τιμαριθμοποίηση κάποιων συμβολέων και επειδή οι περισσότερες δαπάνες που έχουμε είναι στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, οι μειώσει των τιμών κυρίω έχουν γίνει σε άλλες χώρες, στον νότο της Ευρώπης. Μου είπατε να είμαι πολύ συνοπτικό, ίσως δεν ήμουν όσο θα θέλατε, αλλά έκανα ό,τι μπορούσα. Ευχαριστούμε κύριε Γεραματέα, Γραμματέα, ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά τα σχόλια. Προσωπικά θα ήθελα να πω ότι ε, θα σας ζητούσαμε να ε, προγραμματίσετε έτσι ώστε να είμαστε άψογοι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη στιγμή που ζητάμε θυσίες από τους πολίτες μας ή από τα Εθνικά Κοινοβούλια πιστεύω ότι και εμείς ε, θα πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Επόμενη συνεδρίαση στις 16 Μαρτίου. Λίγη συνεδρίαση.